and gentlemen. May I ask take your... Καλησπέρα. Κυρίε και κύριοι, παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε με την έγκριση ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, έχετε κάποια αντίρρηση, ερωτήσεις. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ. Αύριο η ψηφοφορία είναι στις 9. Ε, οι δικοί μου θα δυσκολευτούν να έρθουν. Έχετε καμία αντίρρηση να την κάνουμε 9.30 ή όχι. Ή 10. Mm, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πάντα η ίδια ερώτηση. Ξέρετε ότι προσπαθούμε να μην έχουμε ψηφοφορίες 9. Λόγω ακριβώς ε, του προβλήματος της ε, παρουσίας ε, των βουλευτών. Αλλά στην περίπτωση αυτή έχουμε μόνο μία ψηφοφορία για την στρατηγική των Άλπαιων. Και μετά από αυτό από τις 10, από τις 9.30 έχουμε τον κύριο Γκάιερ εισηγητή από την Επιτροπή Προϋπολογισμού που θα μας πει κάποιες πρώτες απόψεις για τον προϋπολογισμό και μετά συνεχίζουμε με το πρόγραμμα της Επιτροπής. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί χρόνος για αυτή την ψηφοφορία. Γι' αυτό είναι στις 9 η ώρα. So I'll accept that this is acceptable. Okay. Okay. Thank you. Δέχεστε. Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Υπήρξε άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο στο Άμστερνταμ 29 και 30 Μαΐου. Είχε εκπροσωπηθεί η Επιτροπή μας. Η κυρία Βέστφαλιν ήταν στην αντιπροσωπεία. Ο κύριος Όμαζη Αντιπρόεδρος, ο κύριος Φανίστελ Ρόι, ο κύριος Μίλτενμπουργκ και ο κύριος Όλμπριχτ ως επικεφαλής ε, του αστικού intergroup. Η αντιπροσωπεία λοιπόν συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών. Εγώ ως πρόεδρος συμμετείχα στην συζήτηση και Είχα την τιμή να είμαι μαζί με την Επίτροπο την κυρία Κρέτσο και υπενθύμησα το ότι στηρίζουμε ως Κοινοβουλίο την Αστική Πολιτική και τις αλλαγές στο σύμφωνο του Άμστερνταμ που στόχο έχει να στηρίξει το σύμφωνο πόλεων για τις αστικές ζώνες. Επίσης έχουμε και τον ειδικό αστικό απεσταλμένο για την προώθηση καλύτερου συντονισμού των θεμάτων που αφορούν τις αστικές ε, περιοχές. Η παρέμβασή μου βασίστηκε στην έκθεση της Επιτροπής μας και στη θέση της Επιτροπής μας ε, για την αστική ατζέντα και το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Στη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου υπήρχε και άλλη μια συνάντηση στο Άμστερνταμ που οργάνωσε η Επιτροπή των περιφερειών μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον ρόλο των πόλεων και το σύμφωνο του Άμστερνταμ και όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας μας ήταν και σε αυτές τις ε, συζητήσεις. Οπότε, είχαμε ισχυρή εκπροσώπηση κατά την διάρκεια της υπουργικής ε, συνάντησης και νομίζω πως ε, είμαστε ικανοποιημένοι με τις παρουσιάσεις που έγιναν. Τώρα περνάμε στο τρίτο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων ε, με την Επίτροπο, την κυρία Κρετσού, Επίτροπο Αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, σχετικά με το αστικό θέμα θεματολόγιο και την εκ αξιολόγηση Χαίρομαστε που σας καλωσορίζουμε ξανά, κυρία Κρέτσο. Τελευταία φορά τα είπαμε τον Ιανουάριο και χαίρομαι που σας καλωσορίζω και πάλι στην Επιτροπή μας. Μετά από τις αρχικές σας παρατηρήσεις θα δώσω τον λόγο στα μέλη της Επιτροπής για ερωτήσεις και παρατηρήσεις ξεκινώντας από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Επίτροπος πρέπει να φύγει κατά τις 4.30. Αν με χρειάζεται να μείνω. Ναι. Οπότε ο συνήθως δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχετε λοιπόν τον λόγο και μετά θα συνεχίσουμε με την συζήτηση. Χωρίς μικρόφωνο, Επίτροπος. Dear colleagues, uh, uh, good morning. Thank you. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παραστώ σε αυτήν την ε, συνάντηση. Πολύ εύθετη. Τώρα βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι δύο μεγάλων διαδικασιών. Όπως είπε η Πρόεδρος, πριν από δύο εβδομάδες είχαμε πάει στο Αμστερντάμ από κοινού με μια μεγάλη αντιπροσωπεία και την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και είχαμε και την ε, συνεδρίαση την Υπουργική για την ε, ε, ημερήσια διάταξη στο θεματολόγιο των πόλεων, Urban Agenda. Αύριο θα έχω την σύνοδο για την αξιολόγηση στη Σόφια όπου κάποια από τα πρώτα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν για την εκπόστα αξιολόγηση 2007-2013 του προγράμματος εργασιών. Να πω δύο λόγια για αυτά τα, τα γεγονότα και με χαρά θα συνεχίσω το διάλογό μας μετά. Πρώτα με το άτυπο Υπουργικό Συνέδριο στο Άμστερνταμ. Το θεματολόγιο της ατζέντα για τι ε, πόλεις ε, αποτελεί αποκορύφωμα των εργασιών κατά το παρελθόν, ιδιαίτερα με την εμπλοκή και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να δραχθώ τη ευκαιρία να σα ευχαριστήσω για τη διαρκή υποστήριξή σα και ιδέε και προτάσει σα, ε, όπως και για την έκθεση για την αστική διάσταση των πολιτικών της Ένωσης. Το ενεργό έργο σας, η συμμετοχή σας στην διακομματική ομάδα <clears throat> για τις πόλεις Intergroup, Urban Intergroup, είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Αδειμονώ και προσβλέπω στις απόψεις σας για αυτές ε, τις διαδικασίες ε, και τις προτάσεις σας. Η εντύπωσή μου είναι ότι εισερχόμεθα σε μια νέα περίοδο, σε μια νέα εποχή. Και σε σχέση με τόσα αναφέρθηκα στο Άμστερνταμ, η συμφωνία δηλαδή για την ημερήσια διάταξη για τις πόλεις ε, και τα αστικά θέματα πρέπει να θεωρηθεί ένα ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα τη συνθήκη του Μαστρίχ που δημιούργησε την Επιτροπή των Περιφερειών και δημιούργησε και την αρχή της επικουρικότητας με την οποία λειτουργούμε. Φυσικά ήταν ουσιοδός διαφορετικές οι προκλήσεις εκείνης της εποχής από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αλλά και σήμερα όπως και τότε κατά το παρελθόν χρειαζόμαστε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη που θα είναι ικανή να συνενώσει όλες τις δυνάμεις της ε, και το ενεργητό δυναμικό της. Και για τις πόλεις είτε μικρές είτε μεγάλες φυσικά είναι ο πιο στενός ε, σύνδεσμός μας, ε, κρίκος που μας ενώνει με τους πολίτες. Οι πόλεις λοιπόν. Οι πόλεις που βρίσκονται στο προσκήνιο, στο επίκεντρο των απαντήσεων της Ευρώπης για τις προκλήσεις όπως μετανάστευση, κλιματικές αλλαγές είναι ένα ζωντανό πειραματικό εργαστήριο του μέλλοντος η πόλη μας ε- στην Ευρώπη και γι' αυτό πράγματι θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον όλων να δημιουργηθεί αυτή η δυνατότητα διασύνδεσης ε, με τις αστικές εξελίξεις ε, των πόλεων και τις ε, περιοχές υπαίθρου ώστε να υπάρξει μια νέα όθηση για την ολοκλήρωση στην Ευρώπη, ένα νέο άλμα. Και αυτό ακριβώς είναι η πρόταση της Agenda Urban, να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα κονδύλια, καλύτερα να σχεδιάζουμε την ομοθεσία μας και να συμμεριζόμαστε και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας, κυρίως με έναν καινοτόμο τρόπο όπου θα εμπλέκονται οι ουσιώδεις εταίροι. Οι εταιρικέ σχέσει αυτή τη ε, ημερήσια διάταξη ε, για τι πόλει που εμπλέκει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, τι πόλη του εμπλεκόμενου διασφαλίζει ότι δεν θα αφαιθεί ε, εκτό πεδίου δράση κανεί και θα υπάρχει στενή διαβούλευση με τι πόλει επί των θεμάτων αυτών. Από την άλλη πλευρά αλλάζουμε τον τρόπο εργασία μα ώστε να αντανακλάται το πνεύμα τη ημερήσιας διάταξης για τις πόλεις στις εργασίες μας. Βελτιώσαμε τον εσωτερικό συντονισμό και στο πολιτικό και στο τεχνικό επίπεδο. Δεύτερον, δοκιμάζουμε μεθόδους ώστε να μπορέσουμε να, να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για, αυτή, για αυτό το θεματολόγιο και να δημιουργήσουμε μία θηρίδα one-stop shop για τις πόλεις και τα συναφή θέματα. Ε, το έργο μας ξεκίνησε για τις πιλωτικές εταιρικέ σχέσεις για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την ολοκλήρωση ε, και ένταξη των ε, μεταναστών. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η λογική αυτής της ατζέντας θα εντάσσεται στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης διασφαλίζοντας από την άλλη πλευρά ότι θα μπορέσει να απογειωθεί με τις δράσεις αυτές η ημερήσια αυτή διάταξη αυτού του θεματολογίου. Αύριο για την αξιολόγηση θα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να μετρήσουμε τα επιτεύγματα αυτής της πολιτικής και να δούμε πώς θα είναι δυνατόν να, είμαστε, να βελτιώσουμε τα πράγματα στο μέλλον. Θα έχουμε ένα έγγραφο σε επιτροπή που κατ' φθινόπωρο θα δημοσιοποιηθεί, αλλά μπορώ ήδη τα πρώτα μας συμπεράσματα της πρώτης αυτής αξιολόγησης να σας τα αναφέρω. Θεμελιώδες συμπέρασμα. Όλα τα κράτη-μέλη επωφελήθηκαν από την πολιτική συνοχής. Ανάπτυξη, σε μια χώρα που μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις απασχόληση σε άλλες χώρες με βάση τα κονδύλια τα οποία διατίθενται, όπως σας είναι γνωστό, να δείτε πόσες υπηρεσίες και πόσα ωφέλη προέρχονται από ε, εκ των έξω και στις ε, πολιτικές μας αυτές 300 ε, δις ε, συνολικά ευρώ από το 2007-2013 και τα περισσότερα από αυτά στοχοθετημένα έδρασαν στις περιοχές σύγκλησης και συνοχής ώστε να μπορέσει η Ένωση να είναι επιτυχής. Αγαπητοί φίλοι, γι' αυτό θελήσαμε μια πολιτική πανενωσιακή για όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αυθεντική ευρωπαϊκή πολιτική και είμαστε υπερήφανοι για αυτήν ή με την εξπόστα αξιολόγηση όπως καταδεικνύεται την τελευταία φορά τον Ιανουάριο που ήμουν εδώ συζητήσαμε τις επιπτώσεις αυτών των ε, νέων πρωτοβουλειών και στην εξπόστα αξιολόγηση συλλέξαμε τεκμήρια και αποδείξεις για το τι έγινε από το 2007 έως το 2013. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Χάρη στην πολιτική συνοχή, ε, χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν θέσεις απασχόλησης Επίσης 6 εκατομμύρια πολίτες συνδέθηκαν με καθαρά δίκτυα υδροδότησης με καθαρό πόσιμο νερό. Στην πολιτική ολοκλήρωση και ένταξη, ε, χιλιάδε μικρομεσαίε επιχειρήσει μπόρεσαν να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό του, δημιουργώντα ιδανικέ ε, προποθέσει για την διασφάλιση και επέκταση απασχόληση στο μέλλον. Αλλά δεν είναι αυτά όλα και δεν τερματίζουμε εδώ. Με την εξπόστα αξιολόγηση για τι επιπτώσει, μας δίνει την δυνατότητα να λογοδοτούμε για το τι πράττουμε, να διευκολύνουμε τη διαφάνεια και την λογοδοσία προς το κοινό. Ε, επίσης, ε, να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε περιοχές, θέματα όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας προς όφελος των πολιτών. Και όπως γνωρίζετε ήδη, έχουμε στοχεύσει σε μια συζήτηση σε σχέση με τον ορίζοντα 2020 και μετά το 2020. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους ε, και ιδιαίτερα την κυρία Πρόεδρο διότι ξεκινήσατε αυτή τη συζήτηση και έτσι τα πράγματα προωθούνται. Είναι κέρια σημασία οπωσδήποτε να καταφέρουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτά τα δύο μέτωπα. Αφενό να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πολιτική θα είναι αποτελεσματική χάρη στο νέο θεματολόγιο για τις πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου να διασφαλίσουμε ότι η έκθεση θα έχει πραγματικά αντίκρισμα, θα υπάρχει αντίκρισμα των δράσεων αυτών. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα προσβλέπω στις απόψεις σας στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με προτάσεις ε, ή σχόλια ή ε, απόψεις. Ε, πρώτος συντονιστής ο κύριος Βανίστερόη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επιτροπή που ήρθατε για μία ακόμα φορά στην Επιτροπή μας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν γι' αυτό και για τις πληροφορίες που μας δώσατε αλλά προκύπτουν κάποια ερωτήματα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα το σχεδιασμό. Μάθαμε ότι η ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση θα έχει κάποιες, ε, μάλλον έχει κάνει ήδη κάποιες τροποποιήσεις ε, πότε θα έχουμε ε, το χρονοδιάγραμμα πριν τις διακοπές, το Σεπτέμβριο; Επίσης, στην τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια ε, μιλήσαμε για το ΕΦΣΥ και μας δόθηκαν πληροφορίες ότι η Κομισιόν θα αλλάξει τον κανονισμό κοινών διατάξεων όσον αφορά ε, το ε, ΕΦΣΥ έτσι ώστε να, ε, να απλουστεύσει και να διευκολύνει την χρήση κυρίως της πλατφόρμας και των επενδυτικών εργαλείων και θα χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτό ακούσαμε ότι θα έρθει στο Κοινοβούλιο, αλλά πότε θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί αποτελεί δικιά μας νομική αρμοδιότητα. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, κάποιες ημερομηνίε. Πάντα στην ίδια γραμμή, το Κοινοβούλιο θα προωθήσει ε, πρόταση ιδίας πρωτοβουλίας που θα αφορά την σωστή, τον σωστό συνδυασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων και διασφαλίσεων και ε, ε, κυρίως για τα δάνεια, τα grants. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα γιατί θα πρέπει να μας πείτε κι εσείς ποιες είναι οι δικές σας πρωτοβουλίες. Και άλλο ένα σημείο θέλω να θίξω. Μια πρόταση που ε, έφτασε ενώπιον της Επιτροπής μας σχετικά με τα προγράμματα ε, στήριξης ε, των διευθυντικών αλλαγών ή αναδιαρθρώσεων. Έχετε ξεχωρίσει το χρηματικό οικονομικό σκέλος από την τεχνική αρρωγή. Αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς ε, τους στόχους που εμείς έχουμε καθορίσει για την τεχνική ε, αρρωγή. Νομίζω ότι ε, χρειάζεται περισσότερη capacity building στις περιφέρειες. Ωραία μας τα λέτε ε, και όλα είναι ε, πολύ καλά. Έχουμε στοιχεία τα οποία ε, συζητούμε και με άλλες επιτροπές, αλλά θέλουμε και τη δικιά σας άποψη. Και μια τελευταία ερώτηση πιο γενικής φύσεως. Την προηγούμενη φορά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί να συζητήσαμε το ενδεχόμενο η έβδομη έκθεση συνοχής να έρθει νωρίτερα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε για να δουλέψουμε πάνω στους νέους ε, κανονισμούς και ίσως ε, εάν περιμένουμε και την έκθεση να είναι πολύ αργά γιατί το 2019 είναι έτος εκλογών και εσείς αλλάζετε το 20 και ε, κινδυνεύουμε να χάσουμε ακόμα δύο χρόνια. Μήπως θα μπορούσα να έχω λοιπόν από τη δική σας πλευρά έναν σαφή έτσι, χρονικό ορίζοντα, γιατί λέτε ξεκινήσαμε. είναι Πολύ καλό βέβαια που ε, μπορούμε να συζητούμε όλοι μαζί γιατί είναι κάτι κοινό ε, και δεν το συζητάει μόνο το Κοινοβούλιο ή μόνη της η Επομένως, εμείς είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι να κάνουμε το επόμενο ε, βήμα. Μπορείτε να μας δώσετε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύρια Επιτροπέ, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος κυρίας Βεσθάλιν οπωσδήποτε ήθελε να έρθει γιατί το θέμα του συμφώνου του Άμστερνταμ και της αστικής ανάπτυξης να απασχολεί, αλλά δυστυχώ είναι άρρωστη σήμερα και στεναχωριέται και η ίδια. Αλλά, όπως και να έχει, χαίρομαι για το ότι η αστική διάσταση αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας. Θεωρώ πως το χρειαζόμαστε αυτό υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις και η πόλη είναι πολύ σημαντικός εταίρος και πρέπει να τη στηρίξουμε. Και αυτό το οποίο είπατε πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως υπάρχει ακόμα περιθώριο να το ενισχύσουμε και να το βελτιώσουμε και υπάρχει η δυνατότητα στις πόλεις ε, να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Αλλά δυστυχώς στις πόλεις συχνά έχουμε την δυσκολότερη κοινωνική κατάσταση και ίσως οι πόλεις να χρειάζονται την στήριξή μας. Γι' αυτό νομίζω είναι σημαντικό να είναι το θέμα αυτό στην ίδια διάταξη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα, να σας θέσω ένα ερώτημα όσον αφορά την αξιολόγηση της ε, περίοδου 2007-2013. Υπόθηκε ήδη, είμαστε σε μια συζήτηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο και δεν βλέπουν όλοι θετικά την πολιτική συνοχής. Ακούω συχνά ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα λάθη της ε, πολιτικής συνοχής. Μπορείτε εσείς να μας πείτε με δύο-τρία με δύο-τρεις λέξεις, δύο-τρεις προτάσεις ποιες είναι οι χειρότερες εμπειρίες της προηγούμενης ε, προγραμματικής περίοδου και τι πήγε σωστά. τα απλά πράγματα νομίζω πρέπει να μπορούμε να τα μεταφέρουμε για να επηρεάσουμε και τη συζήτηση. Αυτό το οποίο είπε μετά ο Λάμπερτ για τον προγραμματισμό για τους επόμενους μήνες είναι πράγματι σημαντικό και κυρίως μια που οτιδήποτε κάνουμε είτε μιλάμε για τεχνική βοήθεια, το τεχνικό μέσο, η διαδικασία Omnibus είτε η αξιολόγηση δανείων και επιχορηγήσεων, όλα αυτά είναι συζητήσεις όχι μόνο για τα τωρινά θέματα, αλλά και για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και θα ήθελα από σας να μας πείτε κάποια πράγματα πώς το βλέπετε. Θα ήθελα επίση να μου πείτε αν θεωρείτε πως μπορείτε να κανονίσετε τα πάντα με πιστώσεις και με χρηματοπιστωτικά μέσα. Δηλαδή αν έχουμε το εύση και τα υπόλοιπα ταμεία που είναι. Μιλάτε δηλαδή για μια μόχλευση με ιδιωτικό κεφάλαιο. Από πού έρχονται αυτά τα λεφτά. για να προωθήσουμε λέτε το σχέδιο Γιούνκερ. Εγώ θεωρώ πως υπάρχουν κάποια ανοιχτά ερωτήματα τα οποία θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε ως ε, Επιτροπή. Και τώρα να λέμε ότι θα μοιράσουμε παντού επενδυτικά μέσα και αυτό είναι πανάκια, είναι εγγυημένα λάθος αλλά θα ήθελα να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάσιτς, ε, εξο... κυρία Μάσιτς, εξ ονόματος του ΙΣΤΙΑΡ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω σε σχέση με την ανάπτυξη των πόλεων βλέπουμε ότι διοικητικές διεργασίες ε, με τον τρόπο που διοργανώνουμε το έργο μας πολλές φορές επιβαρύνουν τις προσπάθειες ενώ οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές. Ο τρόπος διοργάνωσης δεν δίνει την δυνατότητα να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα και η το πω έτσι, προσέγγιση, πιο ανοιχτή προσέγγιση δεν είναι πάντα εφικτή. Επίσης όσον αφορά για την ανάπτυξη του θεματολογίου των πόλεων, θα έπρεπε να έχουμε παράλληλα και την ανάπτυξη της υπαίθρου ως ε, θέμα που θα παρακολουθούμε εκ παραλίλου. με στόχο οι αστικές περιοχές ε, μια και επηρεάζουν σημαντικά τις περιοχές της υπαίθρου να λαμβάνονται έτσι από κοινού υπόψη θα ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να διασφαλίσει καλά αποτελέσματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό το θεματολόγιο. Uh, κύριε Σφανμελτεμπουργκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε στο Άμστερνταμ την υπογραφή του Συμφώνου του Άμστερνταμ και ήταν θετικό το ότι ήσασταν και εσείς εκεί, αλλά είναι η αρχή της διαδικασίας γιατί τώρα θα πρέπει να βρούμε τις σωστές ε, συνεργασίες για την εφαρμογή του και οι συνεργασίες αυτές ε, είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο εξάμεινο έπαιξε ένα ρόλο και η Ολλανδική Προεδρία βεβαίως ε, χρειάζεται τώρα εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη και υπάρχει όπως είπαμε ευτυχώς η διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την ηγεσία του συναδέλφου Γιάνν Όλμπριχ, η οποία θα πρέπει να αναλάβει δράση για να έχουμε επιπλέον προϋπολογισμό για να λειτουργήσουν αυτές οι συνεργασίες. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν θα βρεθούν τα λεφτά. Έχει μετά σε αυτή την περίπτωση κονδύλια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν αυτές οι συνεργασίες. γιατί βεβαίως εξαρτάται το εάν θα ε, λειτουργήσουν ή όχι ε, όχι μόνο από την βούληση μιας προεδρίας αλλά από την ουσία του χρηματοδότησης. Το δεύτερο ερώτημα έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Βέστφαλε έχει εργαστεί σκληρά για την έκθεση για το αστικό θεματολόγιο και θέλουμε να είμαστε ενήμεροι για το αποτέλεσμα όπως είπα αυτών των συνεργασιών και για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν είναι τόσο σημαντικός ε, στο σύμφωνο του Αμστερνταμ. Μιλάμε συχνά για καλύτερους κανόνες, ε, καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων, αλλά όταν μιλάμε βεβαίω για καλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερους κανόνες θα πρέπει να εμπλέκεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να έχουμε πληροφορίες ε, για το τι γίνεται με αυτές τις ε, συνεργασίες. Ε, το τρίτο θέμα για την ε, αξιολόγηση εκ των υστέρων. Η αξιολόγηση σημαίνει βεβαίως και να αντλούμε και διδάγματα. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλούμε κοιτώντας το τι έχει γίνει εκ των υστέρων και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην αναθεώρηση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ομάρζε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, αλλά και να σας ε, υποβάλω κάποια ερωτήματα. Η Συμφωνία του Άμστερνταμ Γι' αυτό να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, καταδεικνύει την ικανότητα που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανοίξουμε νέες ε, οδούς ε, οι οποίες ε, αργότερα θα ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Γιατί αυτοί που έχουν μνήμη θυμούνται ότι και τα ζητήματα του αστικού θεματολογίου είχαν τεθεί πρώτα στην Επιτροπή Ρέτσι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτήν την ίδια ε, συμφωνία καταδεικνύει την ικανότητα της περιφερειακής ε, πολιτικής ε, να προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις. Και αυτή η ικανότητα προσαρμογής, κατά τη δική μου άποψη, είναι και η αιτία και η προϋπόθεση της συνέχισης της περιφερειακής πολιτικής. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε τα, τα στοιχεία τα οποία αποτελούν την κοινή βάση του συνόλου των πολιτικών ε, που έλκονται από την περιφερειακή πολιτική. Δεν θέλω δηλαδή στο τέλος να βρεθούμε με μία σειρά ε, ξέχωρων στόχων, ξέχωρων μεταξύ τους. Θα πρέπει να έχουμε αυτό τη κοινή βάση ε, την οποία θα διαφυλάξουμε γιατί είναι αυτή η οποία διασφαλίζει την ε, συνοχή και ε, στην έκθεση για την συνοχή θα πρέπει να καταδείξει κάποια στιγμή ότι επετεύχθησαν οι στόχοι γιατί αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνοχή το γεγονός ότι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα οι στόχοι δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε σήμερα αυτή την πολιτική του Θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να σας πω ότι διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την ε, ε, συνέντευξη που έδωσε ο επικεφαλής του γραφείου σας, ο οποίος δεν κρύβει ότι στο Συμβούλιο, όπως και στην Κομισιόν άλλωστε, υπάρχουν ε, ερωτηματικά όσον αφορά το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής μετά το 2020. Και μας μας απασχολεί αυτό ιδιαιτέρως και επομένως τούτη τη χρονιά το 2016 θα πρέπει να την αφιερώσουμε στην ενδυνάμωση των βασικών χαρακτηριστικών της εν λόγω περιφερειακής δηλαδή πολιτικής. Κάτι άλλο που θέλω να πω αφορά τη συζήτηση που είχαμε πριν από μερικές μέρες εδώ στην Επιτροπή μας ε, με τον ε, ε, Επίτροπο Νοβόσκη. Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Επίτροπε, ποια είναι η δικιά σας θέση όσον αφορά τα ζητήματα που τον που το είχαμε θέσει. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι εξεπλάγησαν γιατί για μία ακόμα φορά Αναφερόμαστε στην ε, συνοχή έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν μεταρρυθμίσεις ε, οι οποίες ξεφεύγουν από το πλαίσιο της πολιτικής ε, συνοχής. Ας πούμε, στις διαχρονικές πολιτικές αναφερόμαστε στην μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση με την περιφερειακή πολιτική, αλλά είναι πολύ μακρινή, πρέπει να το ομολογήσουμε. Ευχταίο είναι να έχουμε σύντομα τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί ε, για την απλούστευση. Ε, εμείς λυπούμεθα γιατί η Κομισιόν ε, συνδιαλέγεται με ομάδες εμπειρογνωμόνων και τελικά η Ιερετή ε, στην ουσία ε, διορθώνω με ομάδες εμπειρογνωμόνων οι οποίοι στην ουσία αφαιρούν ε, αρμοδιότητες από τους ερετούς. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο στόχος της απλούστευσης. Είναι η απλούστευση αυτή απαραίτητη έτσι ώστε να προχωρήσουμε στα προγράμματά μας Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση των πολιτικών, νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογούμε έτσι ώστε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να βλέπουμε τι δεν έχει λειτουργήσει καλά, έτσι ώστε να προχωράμε σωστά. Και εδώ θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μια πρόταση, ε, είναι δική μου, δεν της πολιτικής μου ομάδας, ε, που αφορά την ε, δημιουργία μιας αιρεσιμότητας που θα συνδέεται με, τα θεμελιώδη, με τις θεμελιώδες αξίες, ε, με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δυστυχώς ε, είναι ακόμα πολλές οι χώρες οι οποίες καταναλώνουν πολύ τα διαφορετικά ταμεία και που υπολείπονται των ευρωπαϊκών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι έχουμε δεχτεί ε, μακροοικονομικές ε, αιρεσιμότητες ε, γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν ουσιώδες θέμα το θέμα της εξυγίανσης και του χρέους. Εγώ από τη δική μου πλευρά θεωρώ ότι εξίσου σημαντικές και ουσιαστικές είναι και οι αρχές οι οποίες συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είμαστε μια Ευρώπη των αξιών και είναι πραγματικά λυπηρό πολλές χώρες οι οποίες, είναι, ωφελούνται από τα ταμεία και από τους πόρους αυτούς ε, να ε, υπολείπονται όσον αφορά τον σεβασμό αυτών των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που είχατε την ευκαιρία για αυτή τη συζήτηση με την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή σε μια σημαντική φάση του θεματολογίου για τις πόλεις με την εξπόστα και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή έδωσε και τη γνωμοδότησή της ε, για την ε, αναθεώρηση του πολιετούς προγράμματος για το θεματολόγιο των πόλεων. Φυσικά είναι μεγάλη επιτυχία ότι μετά από πολλές συζητήσεις εγκρίθηκε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ένα θετικό ρόλο που διαδραμάτισε από πλευράς του. Εμείς ε, στην ομάδα μου είμαστε κάπως απογοητευμένοι για την έλλειψη, την απουσία του δεσμευτικού ρόλου συμμετοχής των εμπλεκομένων και της κοινωνίας των πολιτών. Εμείς στην πολιτική συνοχή έχουμε την έννοια της εταιρική σχέσης που είναι σημαντικό ζήτημα με δεσμευτική συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, εμπλεκόμενων, μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Και καθότι έχω διαβάσει, καθώς διάβασα το, τη συμφωνία του Άμστερνταμ, η συμμετοχή των εμπλεκόμενων είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Και έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε πάει πιο μακριά και που είχε στην γνωμοδότηση και στην Κοινωνική Επιτροπή και ε, την, είχε δώσει την έννοια της συμμετοχής, υποχρεωτικής συμμετοχής των εταίρων, ερωτώ πώς θα διασφαλίσετε ώστε η εταιρική σχέση αυτή να υλοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο και οι εμπλεκόμενοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δήμοι, κοινότητε, αρχέ, κοινωνικοί εταίροι, μη κυβερνητικέ οργανώσει και κοινωνία των πολιτών υποχρεωτικά, δεσμευτικά να συμμετάσχουν σε αυτή την εταιρική σχέση και να εκπροσωπούνται έτσι δεσμευτικά. Η δεύτερη ερώτησή μου στοχεύει στο πολιετές ε, οικονομικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είχε ήδη εγκρίνει μια γνωμοδότηση από πλευρά και σε σχέση με τους συναδέλφους που προηγούμενα παρενέβησαν και εγώ ενδιαφέρομαι να μάθω σε ποιο βαθμό εσείς τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να δεχθείτε τις ιδέες της Επιτροπής μας. Μια ιδέα θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ και αυτή είναι ότι εμείς είχαμε εκφραστεί για την, κοινωνική, ε, για την πολιτική συνοχή μετά το 2020 και είχαμε τη σκέψη να ξεπεράσουμε το ΑΕΠ ως σημείο αναφοράς. Beyond GDP. Όχι μόνο το, ΑΕΠ να είναι στοιχείο αναφοράς, να μην είναι όμως το μόνο μέσο και στοιχείο αναφοράς και να έχουμε αντίστοιχες, ε, ε, αντίστοιχη εκπόνηση άλλων κριτηρίων όπως κοινωνικών κριτηρίων, καταπολέμησης της φτώχειας, στοιχείων που αφορούν την ανεργία ή και την ισότητα των φύλων. Γνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχουν αντίστοιχε σκέψεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράλληλος προβληματισμός. Είχα αναφέρει ότι σε σχέση με το, την ε, ε, συνέντευξη παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον ε, τις τοποθετήσεις ε, για να ξεπεράσουμε το ΑΕΠ. Δεν θα υποκατασταθεί, δεν είναι αυτή η στόχευση, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί, όχι να υποκατασταθεί, υποκατασταθεί αλλά συμπληρωθεί το ΑΕΠ με άλλα κριτήρια με άλλους ε, γνώμονες ως πύχη για να δούμε πώς προχωράμε. Τελευταία μου ερώτηση, πολύ σύντομα και προσθέτω και εγώ την παρατήρησή μου στην παρατήρηση της Κωνσταντσε Κρέλ προλαλισάσης σε σχέση με το πρόγραμμα Juncker και το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Επενδύσεων. Τι πρόκειται ακριβώς να γίνει σε σχέση με ε, το, τους κινδύνους και ε, κεφαλαίου και πώς ε, μπορεί να καλυφθούν. Δεν δόθηκε ικανοποιητική απάντηση μέχρι τώρα. Ίσως μπορεί να αποσαφινιστεί αυτό. Ποιος θα, ποιος θα είναι ο μύτος της Αριάδνης ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα γιατί πώς ε, βλέπουμε ότι ο κίνδυνος απεμπολείται πλέον σε σχέση με τα κονδύλια αυτά και θα πρέπει λοιπόν εδώ παρακαλώ να δοθεί μια αποσαφήνιση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε την Επίτροπο που ήρθε και σήμερα εδώ. Βράτω με ευκαιρίας της παρουσίας της ε, για να αναφερθώ στον προγραμματισμό 2007-2013 αλλά εάν είναι δυνατόν και ε, για, τον για τη νέα προγραμματική περίοδο. 31 Μαρτίου 2017 λύγει ο προηγούμενος ε, προγραμματισμός, αλλά ε, βάσει των ε, στοιχείων που μας έρχονται από την Επιτροπή Προπολογισμών μπορούμε ήδη να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τα τρία πρώτα χρόνια διαπιστώνουμε στην Ιταλία μεγάλη αύξηση των δαπανών έτσι ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ανεργίας. Θα ήθελα να μας πει ποιο είναι το τμήμα ε, των ε, δαπανών που αφορά αναδρομικές ε, χρήσεις. Επίσης θα μας δώσει ανακράτος συγκεκριμένα στοιχεία έτσι ώστε να δούμε ποια δυσκολία συγκεκριμένη κάθε κράτος αντιμετωπίζει όσον αφορά την απορρόφηση. Επίσης να μας πει εάν είναι δυνατόν στοιχεία τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ολοκληρωθεί ε, ή τα οποία δεν είναι καλη ποιοτητα εάν παρόλα αυτά μπορούν να ενταχθούν ε, στους, τις ε, κεντρικές, στους τελικούς καταλόγους. Θα ήταν δυνατόν η Κομισιόν, ίσως σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Budget, να μας δοθεί, λέω, ένας κατάλογος όλων των πόρων που έχουν δοθεί ανά έργο και ανά χώρα. Επίσης, κάποιες προτάσεις όσον αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ε, οι ε, ρυθμιστικές αρχές, ε, έτσι όπως ορίζονται την 30 Απριλίου του 2016, βλέπουμε σε αυτήν τον κατάλογο μικρό αριθμό ε, ας πούμε 20 ε, διεκδικήσεις αρχές για την ε, Ισπανία με 66 λειτουργικά προγράμματα. Κάτι αντίστοιχο και για την Ιταλία. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ή ότι σε κάθε μία αρχή μπορούν να ανατεθούν περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιο θα είναι το σύνολο των αρχών έτσι ώστε να γνωρίσουμε ε, ανα πάσα στιγμή που βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης. Θα ήταν δυνατόν λοιπόν να έχουμε ένα πίνακα ε, που να μας δίνει τα στοιχεία του συνόλου των αρχών που θα πρέπει οι χώρες να ορίσουν μέχρι την ολοκλήρωση του, της προγραμματικής ε, περίοδου. Μία τελευταία ερώτηση και θα τελειώσω. Σχετίζεται με τις ελεγκτικές λογιστικές αρχές εκτός από τις ε, ε, ρυθμιστικές αρχές, ε, καλό θα ήταν να ξέρουμε και το καθεστώς των αρχών ε, ελέγχου γιατί στην ε, Ιταλία ε, υπάρχουν αρχές οι οποίες είναι ταυτόχρονα και αρχές πιστοποίησης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ακόμα σαφώς ο, η, η αρχή αυτή τότε θα μπορούσε χρησιμοποιώντας το άρθρο 123 να μπλοκαριστεί η διαδικασία διαδικασία ελέγχου. Επομένως, ε, έτσι ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση για την προγραμματική περίοδο μέχρι το 20, ε, ζητούμε την, ε, τον σαφή ορισμό όλων των αρχών ε, των ελεγκτικών ε, και να μας δοθεί από την Κομισιόν ένας κατάλογος με τον συνολικό αριθμό αυτών των εταιριών και των αρχών. Αυτά, αυτές είναι οι ερωτήσεις Να απαντήσετε λοιπόν τώρα σε, αυτήν, σε αυτό το μπλοκ των ερωτήσεων και μετά να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες αυτές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για την δουλειά που έχουμε κάνει. Δεν συμφωνώ ότι δεν ε, υπήρξαν ε, διαβουλεύσεις και βεβαίως η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα είναι μια ευκαιρία να εξετάσουμε πώς λειτουργεί το τρέχον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά ο προϋπολογισμός. Είναι σαφές πως υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ευελιξία και απλοποίηση. Το λέμε εδώ και καιρό. Θα το δούμε αυτό λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως την δουλειά της ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση. Ήδη είχαν κάποιες συστάσεις για το απλοποιημένο κόστος, την ηλεκτρονική συνοχή και επίσης σημαντικό είναι να μεγιστοποιήσουμε τις επενδύσεις στην πολιτική συνοχή. Ε, κοιτάμε λοιπόν τις προτάσεις μας. Και στόχος είναι να έχουμε ένα έγγραφο μετά το καλοκαίρι. Τώρα δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή ημερομηνία, μόλις είμαστε έτοιμοι βεβαίως θα σας ενημερώσουμε. Για την νέα αυτή υπηρεσία, το ΙΑΔΣΕΣ θα έχει στόχο να στήριξη όλα τα κράτη-μέλη κατόπιν ετήματος και η διαθεσιμότητα ε, πρόκειται για κονδύλια της τεχνικής αρχής ε, κατόπιν πρωτοβουλίας της Κομισιόν ε, καθώς και κονδύλια της περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δε αυτά δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα για τα δικά μας κονδύλια της τεχνικής αρχής, της πολιτικής ε, συνοχής. Νομίζω πως υπάρχουν επαρκή κονδύλια για να επιτύχουμε τους ε, στόχους που έχουμε σχεδιάσει. Στον κύριο Φανίστελο απάντησα. Μετά υπήρχαν ερωτήσεις για το αστικό θεματολόγιο και βεβαίως όπως είπα και στην αρχή θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Είναι ένα εργαλείο. Τώρα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο ε, για τα αστικά θέματα, να συνεργαστούμε με τις πόλεις και είμαι πεπισμένη πως το αστικό αυτό θεματολόγιο θα μας δώσει την ευκαιρία να επιτύχουμε τις προτεραιότητες μας μέσω καλύτερης ρύθμισης, χρηματοδότησης και γνώσης και αναμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα εδώ, γιατί μιλήσαμε για συνεργασία. Ε, εδώ πέρα τον ηγετικό ρόλο δεν τον παίζει η Κομισιόν. Είναι μια κοινή προσπάθεια των καρτών μελών, των πόλεων, της Κομισιόν, των ενδιαφερομένων, των ΜΚΟ, των... της και άλλων οργανισμών Πρόκειται λοιπόν για πραγματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Βεβαίω εκτιμώ τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γνωρίζω πως ε, χωρίς εσάς ε, δεν θα ήμασταν εδώ. Βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα στήριζε το αστικό θεματολόγιο, όπως είπα παραδείγματο χάρη μέσω της έκθεσης της κυρίας Βεστφάλτ, για την αστική διάσταση των πολιτικών της Ένωσης μέσω της διακομματικής ομάδας για τα αστικά θέματα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Νομίζω πως μας βοήθησε πάρα πολύ και για το σύμφωνο του Άμστερνταμ και είμαι πεπισμένη πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσφέρει πολλά στο αστικό θεματολόγιο καθώς προσωπεί τις απόψεις των πολιτών. για το χρονοδιάγραμμα τώρα. 24 Ιουνίου αναμένουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί έτσι θα έρθει το αστικό θεματολογίο στην καρδιά των δραστηριοτήτων της Ένωσης και το δεύτερο εξάμενο του έτους προτείνουμε κάποιες επιπλέον συνεργασίες. Είχαμε ήδη ξεκινήσει για την ποιότητα του αέρα, τις ε, εργατικές κατοικίες, τη μετανάστευση κτλ. Και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε και τους 12 θεματικούς στόχους μέχρι το 2017. Θα συνεχίσουμε επίσης ε, να αναζητούμε μεθόδους ε, για να γίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία κατάλληλη για τις πόλεις. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως προετοιμάζουμε και μία ενιαία θηρίδα για να απευθύνονται οι πόλεις και ελπίζουμε ότι έτσι θα έχουμε πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες της Ένωσης. Βεβαίως, Είμαι ευγνώμων και στην ε, Ολλανδική Προεδρία που μας βοήθησε πολύ και προώθησε το αστικό αυτό θεματολόγιο και βεβαίω αναμένω τη συνεργασία και με την Σλοβακική Προεδρία. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε με το τρίο και με τη Μάλτα. Εστιάζουμε λοιπόν στα αστικά ζητήματα, στην αστική σωστικό θεματολόγιο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των πόλεων τον Οκτώβριο και ελπίζουμε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ελπίζουμε λοιπόν να είμαστε σε θέση να δώσουμε και βοήθεια, κάποια ηγεσία και να βοηθήσουμε περιφέρειες, κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή των Περιφερειών. Οπότε, για το ΑΕΠ, βεβαίως νομίζω πως θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε το, το θέμα. Από όσο γνωρίζω το ΑΕΠ είναι το μόνο αναγνωρισμένο κριτήριο αυτή τη στιγμή, αλλά βεβαίως θα λάβουμε υπόψη και άλλους δείκτες, ε, δουλειά, ανεργία, κοινωνικοί δείκτες. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένας νέος ε, δείκτης ε, ευημερίας λέγεται. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το πώς θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά. Για μετά το 2020 Πρέπει βεβαίω να λύσουμε τα διδαγματά μα να βελτιώσουμε την πολιτική. Συμφωνώ μαζί σα ότι έχουμε αυτή την αιρεσιμότητα ex ante που αποτελεί ένα πλαίσιο για καλύτερε επενδύσει, αλλά έχουμε και τις ε, συστάσεις αναχώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα μπορούσαμε να το δούμε σε διάφορες χώρες και συμφωνώ με την άποψή σας πως ε, σε δύσκολους ε, καιρούς πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη και αμοιβαιότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, για τον ε, προγραμματισμό, για να επανέλθω στο ερώτημα του κυρίου Φανίσελρο, η έκθεση η 7η έκθεση προόδου προβλέπεται να γίνει το 2017 και βεβαίω θα προετοιμάσει τις νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν που θα εγκριθούν το 2018. Οπότε είμαι ευγνώμων και προς την Επιτροπή σας γιατί θα αρχίσετε να συγκεντρώνετε κάποιες ιδέες και βεβαίως πρέπει να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και άλλες γιατί κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Και καλό είναι λοιπόν να ακούσουμε κάποιες ιδέες για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε αυτές τις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών, τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. Δεν είναι θέμα μονοπλοποίησης, είναι και θέμα ευελιξίας και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χρειάζονται βιώσιμες επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα να φροντίζουμε η πολιτική μας να μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις και βεβαίως ε, υπάρχει και η σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση, την απόδοση που υπάρχει σε σχέση με την πολιτική μας για τη συνεισφορά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σε σχέση με τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι πρέπει να βελτιωθούμε ακόμα περαιτέρω, ώστε να είναι ακόμα πιο λειτουργική και εύκολη αυτή η πολιτική και οι εποφελούμενοι να μπορέσουν να ελαφρυνθούν και να διευκολυνθούν περισσότερο για τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι ήδη μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σημαντικό να έχουμε τέτοια μέσα για να διασφαλίσουμε τον συντονισμό μεταξύ των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων και του δημιου... της δυναμικού όσον αφορά το Ταμείο Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Και για το θέμα του συνδυασμού κεφαλαίων, φυσικά εργαζόμαστε για αυτό το θέμα με τον κύριο Κατάινεν και θα δοθούν κατευθυντήρες γραμμές πώς είναι δυνατόν να συνδυαστούν τα δικά μας κονδύλια με τα κονδύλια και του προγράμματος Juncker και του στρατηγικού προγράμματος επενδύσεων Μέχρι σήμερα έχουμε ένα μόνο παράδειγμα σε σχέση με τη Γαλλία. Εχθέ άκουσα ότι στην Πρατισλάβα σε σχέση με το ring, το δακτυλίδι της ε, Μπρατισλάβα για το συνδυασμό δηλαδή του αποτελέσματος των κονδυλίων αυτών των ταμείων ιδιαίτερα ως νέο κράτος ε, μέλος χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές, υποστήριξη, αρρωγή να τους συνδράμουμε σε σχέση και με τη δυνατότητα εμπλοκής ιδιωτών επενδυτών που δεν εμπλέκονται τόσο σε αυτό και επίσης και οι τράπεζες δεν μπορούν να προσελκύσουν επαρκώς αρκετούς επενδυτές, ιδιώτες. Σκεφτόμαστε πώς στην ενδιάμεση αναθεώρηση μπορεί να δημιουργηθεί μια δυνατότητα να αποσαφινιστούν περισσότερα τα πράγματα και οι όροι ε, για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Τώρα για την ερώτηση της κυρίας Νταμάτο. Μπορούμε να παράσχουμε ένα κατάλογο των ε, αρχών ε, των κρατών μελών σχετικά. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι μας ανησυχούν πάρα πολλοί καθυστερήσεις και μάλιστα χωρίς τον καθορισμό αυτών των διαχειριστικών αρχών δεν μπορούμε να καταβάλουμε κονδύλια και να κάνουμε πληρωμές. Σε πολλά κράτη-μέλη αυτοί οι διορισμοί δεν έχουν γίνει ακόμα. Και κάθε φορά που συνέρχομαι με υπουργούς, τελευταία φορά συνήθα με τον κύριο Ντεβιτσέντη αναπληρωτή πρωθυπουργό και είναι σαφές ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Επίσης συνάντησα και τον πρόεδρο των, ε, της Νότιας Ιταλίας, των Δήμων Κοινοτήτων του Μεζοτζόρνο της ε, μεσημβρινής Ιταλίας πρέπει να γίνει προσπάθεια να μπορέσουμε ε, σε παράλληλη τροχιά με το άνοιγμα αυτών των δυνατοτήτων να προχωρήσουμε ταχύτατα. Έχουμε ήδη καθυστερήσεις και έχουμε ένα σενάριο αντιμετώπισης ε, των χαμηλής ποιότητας προϊόντων και προσφορών και να μπορέσουμε να δράσουμε ώστε αναδρομικά επισκοπώντας και εξετάζοντας παλαιότερα προγράμματα και σχέδια να βοηθήσουμε με καινοτόμο τρόπο χώρες να μπορέσουν να βελτιώσουν την απορροφητικότητα κονδυλίων. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αναβαθμισμένης ποιότητας, υψηλότερης ε, ποιότητας προγράμματα και σχέδια και πολλές φορές ε, δυσχεραίνονται οι διαδικασίες. Είναι χρονοβόρες, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτόν τον αναστοχασμό, αυτόν τον προβληματισμό ευθύ εξ αρχής τώρα για να βελτιωθούμε στο μέλλον. Νομίζω Αυτά είχα να πω. Αν κάτι ξέχασα μπορώ να επανέλθω. Ευχαριστώ. Θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε στη συνέχεια στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Η κυρία Μαλεύτσε παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, νομίζω ξεκινήσατε, η κυρία Μαλέτιτς, με μια πολύ καλή θετική πρωτοβουλία. Task Force, ομάδα κρούσης για καλύτερη εφαρμογή και υλοποίηση για την περίοδο 2007-2013. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξατε. Είναι πολύ σημαντικό να τα μάθουμε, να ακούσουμε ποια είναι χειροπιαστά αυτά τα αποτελέσματα και πετύχατε σε σχέση με τις δεσμεύσεις σας ε, με τα κονδύλια με τα, ε, με, για τις υποχρεώσεις που είχατε αναλάβει και για το συνεχιζόμενο έργο της ομάδας κρούσης ε, για την περίοδο 2014-2020. Έχετε κάποια στοιχεία αξιολόγησης ε, σε σχέση με τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις μέχρι το 2018 ή και για κάποιες χώρες μέχρι το 2017 έστω. Αυτό ήθελα να πω σε σχέση με το έργο της ε, ομάδας κρούσης Task Force, διότι καλύψατε τις χώρες που είναι πιο αδύναμες ε, σε σχέση με την ε, υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τα διαφορετικά μέσα και την επιλεξιμότητά τους. Έχουμε διοργανώσει κάποιες ακροάσεις. Από ό,τι κατανοούμε από όσους εμπλέκονται στην πρακτική εφαρμογή έχουν πρακτικού χαρακτήρα, χειροπιαστά προβλήματα διαφορετικά μέσα έχουν διαφορετικούς, συνεπάγονται διαφορετικούς κανόνες και οι κρατικοί κανόνες ε, είναι διαφορετικοί. Παραδείγματος χάρη για τον ορίζοντα 2020 και σε σχέση με τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Τι στοχεύετε να πράξετε ώστε να αρθεί, να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η κατάσταση και να αντιμετωπιστούν αυτά τα προσκόμματα, αυτά τα εμπόδια. Τρίτη ερώτηση αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή του ICI και του CB. Κατά πόσον έχουν προχωρήσει αυτά τα νέα μέσα. Έχουμε κάποια καλά παραδείγματα, υποδείγματα σε κάποιες χώρες. Και ίσως μήπως στοχεύετε στο να υποστηρίξετε και κάποιες άλλες χώρες και να διοργανώσετε κάποια ανταλλαγή πείρας, ε, εμπειρίας, ε, πραγματογνωμοσύνης, διότι θα έλεγα ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε την εφαρμογή, την υλοποίηση με, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Ευχαριστώ. Will be from Mr. ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. κύριος Παπαδάκης τώρα. Έχετε τον λόγο κύριε Παπαδάκη. Κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Κρέτσου, ε, η ελληνική κυβέρνηση και ξέρετε έχει σημασία το ότι στην Ελλάδα, στη χώρα μου, η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανη που πρότευσε στην επίδοση της απορρόφησης κονδυλίων φτάνοντας στο 97% της απορρόφησης κονδυλίων ε, της προηγούμενης περίοδου 2007-2013. Δηλώσατε κιόλας υπερήφανη για αυτήν την πολιτική. Η, να κάνουμε έναν απολογισμό για εκείνη την περίοδο τι συνέβη στην Ελλάδα. Από 700.000 άνεργους Έχουμε τώρα 1.500.000 ανέργους. Και αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. 24,2% είναι πολύ ψηλά η ανεργία. Να μην μιλήσουμε ούτε για τα ανεπίσημα στοιχεία, ούτε για, τη, για τους νέους. Επίσης, η, ο κατώτατος μισθός, και, ε, βάζω το, και υπογραμμίζω το θέμα κατώτατος, έπεσε κατά 200 ευρώ. Μοιράζονται οι θέσεις εργασίας, κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας σε 2 και 3 και επί της ουσίας αυτό που έχουμε είναι χειροτέρευση των όρων δουλειάς για τους εργαζόμενους και την ίδια ώρα χρήμα ε, πολύ ζεστό στους επιχειρηματικούς ομίλους που συνάπτουν τα, τις συμφωνίες και με το προηγούμενο πακέτο και με ε, το νέο εταιρικό πακέτο 2014-2020. Η ουσία λοιπόν είναι ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά ταμεία. Άλλο ταμείο είναι αυτό που κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι ε, κερδίζουν και κερδίζουν πάρα πολλά και είναι άλλο το ταμείο και ο λογαριασμός για το λαό, για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται μέσα από την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων η λεγόμενη ανάπτυξη γίνεται στις τάχτες και στα αποκαίδια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Και επειδή συνήθω, επειδή έχω ξαναρωτήσει τέτοιου είδου ερωτήσει, και η απάντησή σα είναι ότι, ξέρετε, αν δεν γινόντουσαν και αυτά, θα ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση. Ε, λοιπόν, η απάντηση είναι, αν δεν, χειρο... αν δεν γινόντουσαν αυτά, θα ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση για του επιχειρηματικού ομίλου. Σίγουρα για το λαό, σε κάθε περίπτωση, είναι ο μόνιμος χαμένος. Και θα ήθελα το σχολείο σας. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κρατσού που έρχεται για μία ακόμα φορά στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω ε, που ήρθε εδώ. Μας είπε ότι θα ότι σύντομα θα έχουμε την αξιολόγηση της προγραμματικής περίοδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να... και για το μέλλον της ε, πολιτικής ε, συνοχής. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε ε, να επιτύχει η πολιτική συνοχή στο μέλλον, αλλά ε, και να έχουμε και μια ισχυρή περιφερειακή ε, πολιτική. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι αυτή η πολιτική ε, καταλαμβάνει μια σημαντική θέση στη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ τα λέω γιατί βεβαίως και η Ουαλία είναι σαφής θετικός δικαιούχος. Ε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Ομάρζη όσον αφορά την απλούστευση. Νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν αν κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, καταλάβαιναν ότι ε, προσπάθεια καταβάλλεται ε, για την πολιτική συνοχή ε, και να ξέρουμε, να ξέρουμε όλοι ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι οι δικαιούχοι, ποια είναι τα μαθήματα που μπορούμε να μάθουμε, ποια λάθη έχουν γίνει και σε τι βελτιώσεις τα λάθη αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν. Να, να ασχοληθούμε δηλαδή, να εμπλακούμε νωρίς στη διαδικασία. Επίσης το θέμα του αστικού θεματολογίου. Ο Επίτροπος Χάνα ε, έβλεπε πολύ θετικά έτσι, το θέμα των πόλεων και της ε, ε, μεταφορά του 5% των κονδυλίων σε πιο μακρινές περιοχές. Ε, δεν ξέρουμε πόσο από αυτά έχουν απορροφηθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί. Ίσως θα πρέπει να μας τα πείτε γιατί ορισμένα προγράμματα βέβαια μόλις ξεκίνησαν ίσως είναι πιο δύσκολο να μας δώσετε στοιχεία. Πάντως καλό θα ήταν στο μέλλον να κάνετε και κάποιους απολογισμούς αλλά και κάποιες προβλέψεις και στο μέλλον καλό θα ήταν Λοιπόν να ξέρουμε τι, ε, ποια είναι τα προγράμματα τα οποία λειτουργήσαν καλά στο παρελθόν. Και νομίζω ότι στα μελλοντικά προγράμματα μια τέτοια διάσταση αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Ρόπκε. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα. Εχθές ε, είχαμε εκπροσώπους της ομάδας Urban και συναντήσαμε και τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης επίσης. Είχαμε μια πολύ γόνιμη συνάντηση και ε, επέτρεψε αρχι, επικεφαλής επιχειρήσεων να θέσουν ερωτήσεις και να κατανοήσουν αυτές τις ε, διεργασίες. Ευχαριστούμε για τέτοιες ευκαιρίες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες Τώρα θα ήθελα να σχολιάσω για τα θέματα της περίοδου 2007-2013 κάποια θέματα. Ήμουν υπεύθυνος για κάποια από τα σχέδια αυτά και μπορώ να πω ότι αυτό που κάναμε είναι ότι είχαμε το ίμιση του χρόνου για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Για την τελευταία περίοδο Μόνο το 2010, κατά τέλη του 2010, μπορέσαμε, μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, γι' αυτό θα έπρεπε να υπήρχαν σαφέστατοι κανόνες. Δύο ή τρία χρόνια για το σχεδιασμό, για προπάσκευη και το υπόλοιπο για την υλοποίηση, την εφαρμογή δεν θα έπρεπε να έχουμε κενές εφρούδες ελπίδες. Τώρα όταν κάνουμε λόγο για το 2014-2020 βλέπουμε ότι οι ίδιοι κανόνες και κανονισμοί εφαρμόζονται. Πρέπει να εγκριθούν πρώτα τα προγράμματα και υστερότερα μετά γενέστερα μόνο μπορούν να υπάρξουν ε, υποβολές προσφορών ε, για την υλοποίηση, εφαρμογή. Στη Λιθουανία για παράδειγμα η κεντρική κυβέρνηση ασκεί πίεση στους δήμους και στις κοινότητες αναφέρεται ότι οι δήμοι και οι κοινότητε δεν χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια, δεν δρούν αρκετά γοργά ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια έγκαιρα, ότι θα έπρεπε να επιταχυνθούν οι διαργασίε, οι διαδικασίε. Μετά γίνονται όμω σφάλματα, συσσωρεύονται σφάλματα και τα πράγματα επιδεινώνονται. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί επίσημα, να καθοριστεί επίσημα ποια περίοδος είναι εκείνη η οποία θα ισχύει για την εφαρμογή, την υλοποίηση και κάνοντας λόγο για τις χώρες ε, όπου υπάρχει κεντροποιημένη κεντρική μορφή σχεδιασμού και εκτέλεσης, για τα βαλτικά κράτη για παράδειγμα, έχουμε θέμα ε, περαιτέρω κατευθυντηρίων, κατευθυντηρίων γραμμών, περαιτέρω λεπτομεριών, δηλαδή η αποτελεσματικότητα στο τέλος τέλος είναι πολύ, σε πολύ χαμηλό επίπεδο με όλους αυτούς τους περιορισμούς. Θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνες διαβούλευσης ε, για να είμαστε πιο επιτυχείς. Δεν σημαίνει αύξηση μόνο επισήμων συνεδριάσεων για ανταλλαγή απόψεων, αλλά θα έπρεπε να αναζητείτε feedback, να αναζητούνται οι απόψεις των εμπλεκομένων. Με αυτόν τον τρόπο, πόλεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν θέματα κλιματικών αλλαγών, αποδοτικότητας ενέργειας, μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα κτλ. θα πρέπει να μπορέσουν να δράσουν πιο αποτελεσματικά. Κατά την προηγούμενη περίοδο δεν αξιολογούσαμε αυτά τα θέματα και θα ήμουν ευγνώμων αν το 2014-2020 θα μπορούσαμε να κάναμε λόγο για την πρόσθετη αξία που θα διασφαλιζόταν. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο παράγοντα, στη συνιστόσα χρόνο και στα χρήματα. Και θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί αυτή η ιδέα να προσεγγίσουμε τις διαφορετικότητα, τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών, σεβόμενοι και προσαρμοζόμενοι σε αυτές τις ε, διαφορές ε, και αυτή τη διαφορετικότητα, ώστε να βελτιωθούν ε, οι επιδόσεις μας. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα Λίλερ για παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα. Τι θα γίνει όμως μετά την περίοδο 2020, εδώ και με την εισαγωγή των ταμείων των κονδυλίων συνοχής για τέτοιου είδους προγράμματα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί σε σχέση με την προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω. Δηλαδή αποτελεσματική χρήση ευθύς... Σας ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ από πλευράς μου λέει η κυρία Μίχελ, συμφωνούμε ότι το νέο θεματολόγιο για τις πόλεις διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, για τον ρόλο ακριβώς των πόλεων. Ένα στόχο που θέλαμε να τον ενδυναμώσουμε, να τον ενισχύσουμε. Η αποτελεσματικότητα όμως εξαρτάται, πιστεύω εγώ, ιδιαίτερα από το πόσο υλοποιείται συγκεκριμένα αυτό το πρόγραμμα και πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια. Γι' αυτό έχω τρεις ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις διατυπώθηκαν, έχω τρεις. Πρώτη ερώτηση. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο πάντα καταβάλαμε προσπάθειες να εμπλακούν περισσότερο οι περιφερειακές αρχές, οι εκπρόσωποι στο περιφερειακό επίπεδο, δήμοι, κοινότητες κτλ. Αναφέρατε ήδη την Επιτροπή των Περιφερειών. Σωστό αυτό και δίκαιο. Ωστόσο όμως προσέξαμε ότι σε κανένα άλλο σημείο σε σχέση με τη συμφωνία, την συνθήκη του Άμστερνταμ δεν αναφέρονται περιφερειακά κοινοβούλια. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τον ρόλο των περιφερειακών κοινοβουλίων, διότι αυτά ακριβώς είτε είναι αστικά κοινοβούλια πόλεων, είτε είναι περιφερειών κοινοβούλια, όποια και να είναι, για την εκπροσώπηση των πολιτών και των συμφερόντων τους διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεύτερη ερώτηση. Ανάπτυξη, αύξηση της αποτελεσματικότητας. Εξαρτάται από τις σαφείς αρμοδιότητες και διαχωριστικές γραμμές και αρμοδιότητες που πρέπει να είναι σαφείς Κάνατε λόγο ότι από πλευρά τη Επιτροπή θα καθορίσετε σαφέστερα με σαφή κριτήρια αυτέ τι διαχωριστικέ γραμμέ για τι αρμοδιότητε. Τρίτη ερώτηση, ίσω απλούστερη. Μέχρι σήμερα όλα τα στοιχεία διατίθενται στα αγγλικά για πληροφόρηση, ενημέρωση. Προβλέπετε εδώ ίσως να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος και να είναι διαθέσιμα και σε περισσότερες γλώσσες για να είναι προσπελάσιμα σε περισσότερους, να διασφαλίζεται η εμπλοκή μεγαλύτερου κοινού. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος ε, Βάλκερ. Ευχαριστώ. Κύριε Βακάσερ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εμείς προσθέτουμε τη φωνή μας ε, στην έκφραση ευχαριστειών προς την κυρία Επίτροπο, διότι αυτό το χρόνο τον συμμερίζεται μαζί μας, ε, τον επενδύσεως, ώστε να είναι μαζί μας για να εξεταστούν θέματα μεγάλης σπουδαιότητας σε σχέση με την περιφερική ανάπτυξη. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης ε, και την Ολλανδική Προεδρία και όλα τα θεσμικά όργανα που ενεπλάκησαν στην υπογραφή, προς υπογραφή της ε, Συμφωνίας του Άμστερνταμ για το αστικό θεματολόγιο, για το θεματολόγιο των πόλεων, την, την ανάπτυξη των πόλεων τον προηγούμενο Μάιο. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει ένα ρόλο σημαντικό στην υλοποίηση όλων αυτών όπως είναι επίσης σημαντική η συνιστόσα των πόλεων στις ευρωπαϊκές πολιτικές και η ενίσχυση του συντονισμού και των επιπτώσεων στον τομέα των πόλεων και να δούμε να ανοίξει μια θηρίδα μία και ενιαία ε, για τα θέματα της ανάπτυξης των πόλεων. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει εκμεταλλευομένη της ευκαιρίας της αναθεώρησης, ενδιάμεσης αναθεώρησης τα στοιχεία που αφορούν την συλλεγήσα εμπειρία με τα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων σε σχέση με τη στρατηγική 2020. Επίσης θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για την αξιολόγηση ex post σε σχέση με το 2007-2013. Παρότι βοήθησε η πολιτική συνοχή στη μείωση των περιφερειακών διαφορών, πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιπτώσεις δεν είναι καθόλου ενιαίες. Κάθε άλλο μάλιστα. Ε, σε σχέση με την πολιτική συνοχή δεν μπορεί να ταυτοποιείται απλά και μόνο εξετάζοντας κάποια στοιχεία για το ΑΕΠ και άλλες, άλλους οικονομικούς συντελεστές. Και γι' αυτό οι δείκτες ε, του ΑΕΠ ανακεφαλή δηλαδή πρέπει να συμπληρώνονται με άλλους δείκτες για να μπορούμε να υλοποιήσουμε μια αξιολόγηση πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική. Δείκτες όπως την απασχόληση, τη φτώχεια όπου αναφέρθηκε σε αυτά τα θέματα η κυρία Επίτροπος. Τέλος και ολοκληρώνω η απλούστευση, η απλοποίηση της πολιτικής συνοχής είναι χωρίς αμφιβολία αναγκαία και πρέπει να επιτευχθεί. Και ως προς αυτό έχει σημασία κλειδιού να ενισχύσουμε το διοικητικό δυναμικό και τη διαφάνεια. Ταυτόχρονα με τη διασφάλιση επαρκούς επίπεδου αυτοδυναμίας χρηματοοικονομικής για να είμαστε αποτελεσματικοί. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται η ανάπτυξη του διοικητικού δυναμικού και να πρικοδοτήσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την πολιτική συνοχή. Για όλα αυτά που προανέφερα θα θέλαμε να γνωρίζουμε, κυρία Επίτροπε, Πώς ε, θεωρείτε ότι μπορείτε να βοηθήσετε τις ε, αρχές των πόλεων για να υπάρχει πιο συστηματική εργασία και πιο αποτελεσματική δουλειά. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις ε, θα αναλάβετε σε σχέση με το να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση και απλούστευση σε σχέση με τα θέματα των πόλεων. Και τέλος, με ποιο τρόπο θα αυξήσετε τις συνέργειες και τον αποτελεσματικό, την αποτελεσματική χρήση των μέσων και εργαλείων ως όπλων σε σχέση με τις συμφωνία δήμων, δημάρχων κτλ. Ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Έχετε χρόνο λοιπόν να απαντήσετε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μου υποβάλατε. I think I forgot to respond to... Νομίζω ότι πριν ε, ξέχασα να απαντήσω στην Κωνσταντσε. Κοιτάξτε, εγώ δεν, δεν θέλω να λέω ονόματα. Αυτό το name and shame δεν με βρίσκει σύμφωνη. Ε, ε, υπάρχουν περιπτώσεις καλής καλών εμπειριών, αλλά υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι αρνητικές ε, και δεν μπορούν να επαναληφθούν. Και όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε ε, ε, αργοπορίες σε πολλές χώρες. Έδωσα κάποια στοιχεία για την περίοδο 7-13 και ξέρετε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες δούλεψαν καλά ή μάλλον είχαν καλή, καλές επιδόσεις αλλά βεβαίως ταυτόχρονα πρέπει από τις εμπειρίες μας να μάθουμε. Κυρία Μάλετιτς. Task Force για καλύτερη υλοποίηση. Ξέρετε ότι την πρώτη φορά που ήρθα στην Επιτροπή ανακάλυψα ότι κάποιες χώρες ε, είχαν συγκεκριμένα έτσι, προβλήματα όπως ε, χώρες ε, καινούριε Βουλγαρία, Κροατία αλλά και Ιταλία, Σλοβενία, Ουγγαρία και αποφάσισα λοιπόν ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην Task Force για την καλύτερη υλοποίηση. Ήταν πολύ καλή σκέψη ε, είχαμε 20 αλλά μπορεί και 30 ε, συναντήσεις. Μάλιστα το 2015 καταφέραμε να μην χάσουμε χρήματα σε μερικές χώρες. Ας πούμε στην Ιταλία όταν ανέλαβα ε, οι υπηρεσίες μου, μου είπαν ότι δεν θα ήταν δυνατόν να κλείσουν μέχρι το τέλος του χρόνου τα επιχειρησιακά προγράμματα. Πήγα στη Μεσημβρινή Ιταλία τρεις φορές, κυρίως Καλαβρία, Καμπανία, Σικελία, που που παρουσιάζονταν οι πολύ μεγάλες ε, ε, καθυστερήσεις ε, και με αυτήν την Task Force για την καλύτερη υλοποίηση καταφέραμε να κλείσουμε τα προγράμματα. Συνεργαστήκαμε με τις εθνικές αρχές και μέσω ε, αυτής της Task Force ε, μπορούμε να δείξουμε ισχυρή στήριξη ε, προς τις χώρες αυτές και αυτό τελικά εστέφθη από, επιτυχία. Τώρα θα αξιολογήσουμε την δουλειά αυτής της Task Force. Ίσως το δεύτερο τμήμα του 2016 να έχουμε την ε, δυνατότητα ε, να καταλήξουμε σε κάποιες συγκεκριμένες ε, ιδέες και προτάσεις όσον αφορά την Κροατία που είναι και το νεότερο μέρος, μέλος. Συγγνώμη. Θα συνεχίσουμε και μέχρι το τέλος του 2016, ίσως και μετά, να παράσχουμε συγκεκριμένη στήριξη βοήθεια στη χώρα. Ε, και ζήτησα από τις υπηρεσίες μου ε, να συστήσουν μια ειδική ομάδα ε, για την Κροατία, έτσι ώστε να στηρίξουν την Κροατία με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά, σημαντικό, όσον αφορά τις ολοκληρωμένες επενδύσεις. Κοιτάξτε, εγώ ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρο της Περιφέρειας Μούρθια ε, και μου παρουσίασαν κάποια προγράμματα ε, για την ολοκληρωμένη περιφέρεια η οποία ε, περιλαμβάνει πέντε πόλεις και στα πλαίσια αυτής της επένδυσης μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συνολική υλοποίηση και με τον τρόπο αυτό μπορούμε και να προχωρήσουμε με πιο επιτεχημένο ρυθμό. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνοδεύει, βοηθάει ε, τις χώρες, τις βοηθάει να ξεπεράσουν τις ε, δυσκολίες της και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό στα ITI μπορούμε να έχουμε πρόοδο. Για την Ελλάδα τώρα. Για την Ελλάδα λοιπόν. Τι μπορώ να σας πω. Μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας ε, ότι η Ελλάδα διανύει δύσκολη κατάσταση. Είχατε την οικονομική κρίση, είχατε τη μεγαλύτερη κρίση μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσθέθηκε ε, και το προσφυγικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξέρετε ότι ήταν πάντα στο πλευρό της Ελλάδας για να βοηθήσουν την Ελλάδα ε, και ε, σας ζήτησα και το ψηφίσατε στην Επιτροπή σας ε, μια επιπλέον βοήθεια για την Ελλάδα. Επομένως αυτό, αυτή η απορρόφηση ε, του 97% ε, αφορά την συγχρηματοδότηση. Μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας βεβαίως ότι η κατάσταση όσον αφορά την ανεργία ε, κλπ. είναι ιδιαίτερα χαλεπή Απ' την άλλη πλευρά, ε, φανταστείτε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στην Ελλάδα ε, αν δεν είχε υπάρξει αυτή η πολιτική ε, συνοχής, ε, γιατί πάνω από 100 εκατομμύρια δις ευρώ είναι η συνολική, η συνολική χρηματοδότηση, δηλαδή από την οποία έχει ευεργετηθεί η Ελλάδα. Υπήρξε και σε έργα υποδοχή υποδομής, ε, ε, δρόμους, μετρό στην Αθήνα, σχολεία, τώρα μετρό στη Θεσσαλονίκη, ε, όλα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα είχαν γίνει ενδεχομένως εάν δεν έχει υπάρξει αυτό ε, αν δεν είχε υπάρξει αυτή η ε, χρηματοδότηση. Ε, συμμετέχουμε επίσης, εκτό από το μετρό της Θεσσαλονίκη και στη διαχείριση απορριμμάτων της Αθήνας. Είναι μοιρασμένη η ευθύνη για το ότι συμβαίνει στην χώρα. Εγώ μπορώ να πω ότι χαίρομαι, είμαι περήφανη γιατί καταφέραμε να προχωρήσουμε στη συγχρηματοδότηση, να αλλάξουμε τον κανονισμό ειδικά για την Ελλάδα και να σας πω ότι από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα η Ελλάδα έχει λάβει πάνω από δύο δις που δεν έχουν λάβει άλλες χώρες. Επομένως, βοηθούμε την Ελλάδα και την έχουμε βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισε. Είναι σημαντικό λοιπόν να ε, έχουμε μοιρασμένη ε, ευθύνη και πραγματικά εμείς το δικό μας το κομμάτι ε, το ε, καλύψαμε. Ε, ε, θα πρέπει να σας πω ότι κατανοούμε την κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Βοηθήσαμε και όσον αφορά την προσφυγική κρίση, όπως βοηθήσαμε και την Ιταλία για το ίδιο ζήτημα. Απ' την άλλη πλευρά, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει και η δυνατότητα απορρόφησης όλων των κονδυλίων π.χ. για την προσφυγική κρίση. Ε, Ντύρκ, αν δεν σε ξαναδώ μέχρι το τέλος του ε, μήνα, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Μετά την διάσκεψη της ε, Σόφιας ε, που θα γίνει σε μερικές ε, μέρες νομίζω ότι θα είμαι σε θέση να σας δώσω και κάποιες γραπτές πληροφορίες και μετά από το τέλος του καλοκαιριού βεβαίως θα έχουμε και την κανονική, τα κανονικά αποτελέσματα της αξιολόγηση. Σύμφωνο μαζί σας ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε κατά την άποψή μου ε, αυτή είναι μια ιδιαίτερος ορατή, αν όχι η πλέον ορατή ε, ενωσιακή πολιτική. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πραγματικά γιατί είναι ε, αυτή η οποία δέχεται, αυτή η πολιτική η οποία δέχεται για τις περισσότερες επιθέσεις. Έρχεστε από περιφέρειες και ξέρετε την κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία περιφέρεια η οποία να μην ωφελείται από κάποιο σκέλος της της ε, περιφερειακής ε, πολιτικής ή της ε, πολιτικής συνοχής. Έχουμε πολλούς επικεφαλείς περιφερειών που μας ζητούν να μην αλλάξουμε αυτή την πολιτική γιατί διαφορετικά φοβούνται ότι δεν θα έχουν άλλη δυνατότητα χρηματοδότησης όσον αφορά το την Urban Agenda. 15 δις θα διαχειρίζονται οι πόλεις άμεσα τα επόμενα χρόνια. Και αυτό βεβαίω είναι μεγάλη ευθύνη. Ε, επομένως θα πρέπει να, έχουμε, να κάνουμε την προσπάθεια να καταβάλουμε όλη την προσπάθεια για καλύτερη ε, συνεργασία και επικοινωνία και η κυρία Βάνα το ανέφερε αυτό, ε, καλή επικοινωνία έτσι ώστε ε, να έχουν όλες οι πόλεις την δυνατότητα να διαχειριστούν καλά το αστικό θεματολόγιο, τις άμεσες επενδύσεις κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι σημαντικό να μιλάμε με, τους, με τα Υπουργεία αλλά και με τις τοπικές αρχές. και αυτό, αυτή η καλή επικοινωνία ε, θα έχει θετικά αποτελέσματα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί ε, ε, και τα κοινοβούλια μάλλον τα τοπικά ε, ήρθα σε επαφή ε, ας πούμε και με την, ε, το τοπικό κοινοβούλιο της Βαβαρίας και γενικώ πάντα όταν επισκέπτομαι περιφέρειες προσπαθώ να επισκεφτώ και τις, τα κοινοβούλια τους. Εν πάση περιπτώσει να σας πω ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να αποφασίσουν μόνες τους ε, να εμπλεκούν. Να εμπλακούν. Και εμείς ε, θέλουμε επαφή, τους καλούμε και τους ε, υπευθύνους, τους επικεφαλείς των περιφερειών. Περίοδος 7-13 επανέρχομαι και λέω ότι έχετε δίκιο. Ε, εγκρίναμε τα προγράμματα ένα χρόνο πριν και σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, δεν έχουμε ακόμα ορισμένη δεν, δεν έχει, και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμα οριστεί η ρυθμιστική αρχή. Αυτό δεν είναι καλό. Κατανοώ βεβαίως ότι κάποιες χώρες είναι πιο καινούριες, αλλά άλλες είχαν 7 χρόνια εμπειρία. Ε, και νομίζω ότι κάτι πρέπει να μάθουμε από αυτά τα 7 χρόνια ή κάτι ε, έπρεπε να έχουν μάθει οι χώρες αυτές. Και άλλωστε στόχος αυτής της πολιτικής είναι η μείωση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών. Ε, ευελπιστώ ότι το 2016 δεν θα είναι χαμένη χρονιά για τα κρατημέλη, γιατί σε πολλές χώρες μέλη έχουμε απορρόφηση της τάξης του 0,1, 0,2 κτλ. Η κυρία Μίχελς επίσης ε, αναφέρθηκε στα τοπικά κοινοβούλια ε, και στο αστικό θεματολόγιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τα υπενθυμίζουμε αυτά. Κύριε Βαρκάρτσελ, ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Στο αστικό θεματολόγιο εμείς αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία. Δίνουμε επίσης ε, ε, τον, ε, τη δυνατότητα σε όλους να έχουν το ίδιο βάρος μέσα σε εταιρικέ σχέσεις με πραγματογνωμοσύνες κλπ. Στην Κομισιόν εμείς έχουμε αναλάβει έτσι κάποιο συντονισμό όσον αφορά ε, αστικά θέματα και βεβαίως η Κομισιόν ε, θα εμπλακεί στην υλοποίηση όλων των ε, σχεδίων δράσης που θα πρέπει να υποβληθούν στην Κομισιόν, όπως θα πρέπει να υποβάλλονται και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο περιοδικές τακτικές αναφορές ε, όσον αφορά ε, την εξέλιξη. Εμείς ε, είμαστε ανοιχτοί για βοήθεια, για έγγραφα, για να παράσχουμε προσανατολισμό, τεχνική αρρωγή να βοηθήσουμε στη διασύνδεση με άλλα Ινστιτούτα ή με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως οι Ηνωμένα Έθνη. και ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα προχωρήσει καλά αυτό το αστικό θεματολόγιο. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που με αφιερώσατε, ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Θα είμαι πάντα ε, στην διάθεσή σας και αμέσως μετά το καλοκαίρι θα ξαναέρθω. Ευχαριστούμε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας χαρίσατε, για τις απαντήσεις, τις πληροφορίες. Θα ξανασυναντηθούμε ουσιαστικά το Σεπτέμβριο, μετά τις ερηνες διακοπές. Όμως αύριο και μεθαύριο πραγματικά υπάρχει μια μεγάλων διαστάσεων σύνοδος στην Σόφια για την αξιολόγηση εξ Και στη συνέχεια από αυτή την σύνοδο θα παρουσιαστούν όλα τα χρήσιμα στοιχεία. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ Επίτροπε. Ε, τώρα κυρίες και κύριοι μπορούμε να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. The next... Το επόμενο... Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη για το απόγευμα, το σημερινό απόγευμα, είναι μια δημόσια ακρόαση, όπως προβλέπετε, για την αξιολόγηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαθωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Αυτή η ακρόαση συμπληρώνει την προπαρασκευή για την έκθεση υλοποίηση πάνω στο ίδιο θέμα που συντάχθηκε από τον κύριο Φανίστερ Ρόι. Το πρόγραμμα για την ακρόαση σας έχει ξεχωριστά διανεμηθεί και για να σας δώσω κάποιες πληροφορίες πώς θα διοργανώσουμε αυτή την ακρόαση Πρώτα θα λάβει τον λόγο ένας, ένας όσοι έχουν προσκληθεί για 10 λεπτά ο καθένας. Ήδη παρευρίσκονται. Μετά θα πάρουν τον λόγο τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για ερωτήσεις και σχόλια και ε, η Επιτροπή αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση δίνοντας τον λόγο στον εισηγητή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. και με τις παρατηρήσεις ναι, μάλιστα, του εισηγητού της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για να υπενθυμίσω ότι εμείς είμαστε συνδεδεμένοι. Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι συνδεδεμένη η Επιτροπή σύμφωνα με, τον, με το άρθρο 54. Καλωσορίζουμε τον κύριο Πυρίνσκι στη συνεδρίασή μας. Και θα έλεγα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τις συζητήσεις μας και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ρον Βαν Ράκ, επικεφαλής προγράμματος για τις ευκαιρίες από την Ολλανδία. Έχετε τον λόγο κύριε, παρακαλώ. Thank you. Thank you for... Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε να κάνω κάποια σχόλια για την διαδικασία των ε, διαπραγματεύσεων και το τι κάναμε για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εγώ είμαι επικεφαλής ε, της ε, διαχειριστικής αρχής της Δυτικής Ολλανδίας, όπου ζει περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας. Εκεί βρίσκεται το Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ αρκετές ε, καινοτομίες, αλλά είναι αρκετά μικρό το πρόγραμμα. Έχουμε 189 εκατομμύρια στο ΕΤΠΑ, τα οποία μειώθηκαν ε, σε σχέση με την περίοδο 2007-2013. Σκοπεύουμε λοιπόν ιδιαίτερα να προωθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, χαμηλού άνθρακα και βεβαίως ε, το ζήτημα των προσόντων στην ε, αγορά εργασίας, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ακριβώς τα προσόντα των εργαζομένων. Θα αναφερθώ λίγο στις πέντε πτυχές των νέων κατευθύνσεων που έχουν δοθεί για τις διαπραγματεύσεις 2014-2020. Ε, Άκουσα κάποιες σκέψεις ήδη από τους ε, βουλευτές και θα δείτε ότι μας απασχολούν αυτά και στην πράξη. Αν δούμε τις συστάσεις ε, ανά χώρα, θεωρώ πως συνδυάζονται αυτά με τους θεματικούς στόχους για να έχουμε αποτελεσματικά προγράμματα. Ειδικά οι διαρθρωτικές συστάσεις ήταν πάρα πολύ χρήσιμες για να εστιάσουμε περισσότερο στην αποτελεσματικότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από το δικό μου πρόγραμμα. Είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη όταν μιλάμε για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και βασική έρευνα, αλλά δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να αξιοποιήσουμε πρακτικά αυτά τα ζητήματα και η σύσταση ήταν ακριβώς να προχωρήσουμε περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή τους ε, και επιλέγουμε ακριβώς προγράμματα που ε, προχωράνε παρακάτω στην αλυσίδα της ε, καινοτομίας. Οπότε ήταν μια σωστή κατεύθυνση. Είμαι κάπως πιο αρνητικός όσον αφορά την αιρεσιμότητα ex ante. Νομίζω ότι γενικά υπήρχαν πολλοί όροι, οι οποίοι δεν ήταν πολύ αποτελεσματικοί, ειδικά για δύο λόγους. Οι βασικοί φορείς οι οποίοι πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το θέμα δεν είναι οι ίδιοι στην χώρα μας ε, και στις άλλες χώρες νομίζω. Ε, οι ίδιοι οι οποίοι εφαρμόζουν τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Είχαμε λοιπόν αρκετές ε, καθυστερήσεις. Οπότε είχε λίγο το αντίθετο αποτέλεσμα λόγω ακριβώς αυτής της ρεσιμότητας εκ των προτέρων και βεβαίως δεν υπήρχε πάντα και μια αναλογικότητα με τα ποσά, τα κονδύλια των προγραμμάτων. Οπότε αυτή η εξάντε ερεσιμότητα μας βρίσκει λίγο αντίθετους τώρα. Τα διδάγματα τα οποία αντλήσαμε. Η έξυπνη εξειδίκευση εστίασε στην οικονομική ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής. Νομίζω επίσης πως μερικές φορές ήδη ισχυρε πολιτικές για την καινοτομία στο περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ε, εξαντερεσιμότητα αντί για μια νέα πολιτική. Αυτή είναι μια βελτίωση που νομίζω πρέπει να επέλθει όταν υπάρχει ήδη μια καλή πολιτική καινοτομία ε, και δεν χρειάζεται μια έξυπνη πολιτική σε Θεωρώ λοιπόν πως έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια έξυπνη εξειδίκευση και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η δικιά μου λοιπόν η συμβουλή είναι η εξή Να έχουμε περιορισμένη και αναλογική ε, στρατηγική η οποία θα πηγαίνει προς μια έξυπνη εξειδικευσή. Μια πρόταση κάπως πιο επαναστατική να βρούμε μια αιρεσιμότητα εκ των προτέρων για να μην ε, βάζουμε ό,τι θέλουμε ε, στο επίπεδο του προγράμματος, να προσπαθήσουμε δηλαδή να περιορίσουμε κάπως την ε, ενέργεια που θα αφιερώσουν εθνικές και τοπικές αρχές για να εφαρμόσουν τα προγράμματα. Μετά περνάμε στο επόμενο. για την ε, θεματική εστίαση. Πάρα πολύ σημαντικό θεωρούμε για να βρούμε και κάποια αποτελέσματα, δηλαδή δεν είχαμε έναν ευρύτατο στόχο, αλλά έπρεπε ε, να επιμείνουμε στα συγκεκριμένα προβλήματα και στις θεματικές επιλογές που είχαν γίνει. Τα διδάγματα που αντλήσαμε ήταν πως οι ε, διαπραγματεύσει ήταν ίσως κάπως πολύ τεχνικές, ε, δηλαδή τι εννοώ, κάποιες δραστηριότητες όταν βγαίνονται ε, κάποιες θεματικές επιλογές ε, μας τις απαγόρευε η Κομισιόν, μας έλεγε ότι δεν ταιριάζουν την χύψη θεματική επιλογή αλλά νομίζω πως θα έπρεπε να δώσουμε βάρος στην συνεισφορά του θεματικού στόχου και όχι στο ποιες ε, δραστηριότητες θα πρέπει να γίνονται. Καμιά φορά μια δραστηριότητα η οποία δεν θεωρείται χρήσιμη σε ένα θεματικό στόχο μπορεί να δοκιμαστεί και αυτή. Θα προτιμούσα λοιπόν οι συζητήσεις να αφορούσαν περισσότερο το γιατί έγιναν κάποιες επιλογές ε, και όχι το ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες επιτρέπονται και ποιες όχι. Μετά, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Νομίζω είχαμε επιτύχει στην περίοδο 2014-2020 και λόγω του κώδικα συμπεριφοράς να έχουμε περισσότερους ενδιαφερόμενους να, να προετοιμάσουμε τις, ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα και έτσι καταφέραμε να έχουμε περισσότερους ε, συμμετέχοντες ε, και από ένα ευρύτερο φάσμα. Και βέβαια είναι δύσκολο ακόμα να υπάρξει κάποια βελτίωση γιατί αφενός ε, θα θέλαμε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν κάποιο ρόλο και στην επιλογή των έργων. Από την άλλη υπάρχει το θέμα της ανεξαρτησίας εκεί πέρα. Οπότε βλέπουμε τώρα πως ο ρόλος τους είναι κάπως πιο περιορισμένος από ό,τι περιμέναμε ίσως. Οπότε πρέπει να βρούμε κάποια μέσα για να έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία θα ανταποκρίνονται στην ζήτηση για να κάνουν ε, οι ενδιαφερόμενοι αυτό το οποίο χρειάζεται από τις εταιρείε και τα διάφορα ερευνητικά ιδρύματα σε καθημερινή βάση. Επίσης για την πολυετή, την, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχουμε κάποιες επιφυλάξεις Στη μισή ώρα που σας άκουσα αναφέρθηκε για το ΕΦΣΙ, το καινούργιο ταμείο και τα διαρθρωτικά ταμεία. Βλέπουμε πως δεν υπάρχει ο ίδιος μηχανισμός και οι ίδιοι κανόνες, οπότε είναι δύσκολο να υπάρχει κάποια συνέργεια. Επίσης, αν δούμε την διαχείριση των δύο μέσων είναι τελείως διαφορετική και οι περιφερειακές ε, κυβερνήσεις ε, ε, μάλλον δεν έχουν και αυτές την δυνατότητα να ε, εμπλακούν. Μετά είχαμε μια περισσότερη μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα των αποτελεσμάτων. Τώρα είναι κάπως νωρίς να κρίνουμε εάν ε, είχαμε επιτυχία ή όχι, γιατί είναι δύσκολο να δούμε εάν οι δείκτες απόδοσης οι οποίοι θα μετρηθούν για πρώτη φορά το 2018 ε, και θα ανταμυθούν ή όχι αναλόγως με κάποια επιπλέον κονδύλια. Αν λοιπόν ε, οι δείκτες αυτοί ήταν επιτυχημένοι. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια αξιολόγηση εάν δηλαδή η λογοδοσία είναι εύκολη και αξιόπιστη για να πούμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερο κομμάτι ή εάν θα πρέπει να γίνει κάτι στην επόμενη εξευρήση. Αλλά νομίζω ότι γενικά είναι ένα καλό μέσο. Επίσης, βλέπουμε πως ε, στις διαπραγματεύσεις προέκυψε ότι θα πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση στα κίνητρα και στην λογική αντί για τα τεχνικά ζητήματα που μας απασχόλησαν πολύ περισσότερο από την επιλογή των δικτών. Οπότε από την δικιά σας την σκοπιά των διαπραγματεύσεων ε, θα ήθελα όπως είπα αυτές να είναι κάπως λιγότερο τεχνικές ε, και να κοιτάνε κάπως περισσότερο την λογική που υπάρχει πίσω από τα προγράμματα. Μετά Αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμή είναι πάρα πολύ ε, καλά. Στο ΕΤΠΑ που είναι η δικιά μου ειδικότητα είδαμε μεγάλη μείωση, μεγάλη απλοποίηση, μεγάλη μείωση του διοικητικού βάρους. Ένα άλλο μειονέκτημα που έχουμε τώρα είναι ότι έχουμε τέσσερις φορές περισσότερες σελίδες ε, κανονισμών σε σχέση με το 2007-2013. Έχουμε πολλές ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση και, και τα κείμενα είναι πολύ πιο μακροσκελή. Βεβαίως, ε, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν είναι απλά ή ότι είναι χειρότερα, αλλά συχνά πρόθεται η χρήση διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων. Υπάρχουν πολλέ υποχρεώσει, πολλοί αυστηροί κανόνε, οπότε έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε για να γίνουν πιο ευέλικτοι και να συνδυάζονται και με του εθνικού πόρου ε, και το Ταμείο Juncker. Και συμφωνήσαμε βεβαίω ε, να αυξηθεί η συμμετοχή μας από το 10% στο 40% 100 ε, αλλά όπως είπαμε είναι δύσκολο να ε, ανταποκριθούμε σε όλους τους κανονισμούς. Και επίσης ένα πρόβλημα είναι ότι οι κανονισμοί αλλάζουν, δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν έχουμε ακόμα όλες τις ε, ερμηνείες από την Κομισιόν και πρέπει να περιμένουμε στις τελευταίες αυτές πράξεις κατεξιοδότηση και δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα και όλα αυτά βεβαίως ε, δημιουργούν καθυστέρηση γιατί πρέπει να υπάρχει νομική βεβαιότητα εκ των προτέρων ε, στους δικαιούχους για το τι ε, θα πρέπει να περιμένουν και τι πρέπει να κάνουν με αυτά τα έργα. Για την συνέργεια. Τώρα έχει υπάρξει κάποια βελτίωση. Έχουμε συνδυασμούς μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ΕΤΠΑ ε, κάτι το οποίο διευκολύνει και η νομοθεσία αλλά τα ταμεία βεβαίως είναι ακόμα χωριστά όσον αφορά την λογοδοσία και οι κανονισμοί δεν είναι ίδιοι οπότε νομίζω πως μπορούν να γίνουν κάποια βήματα ακόμα για να ενισχυθούν οι συνέργειες και μετά το άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί χρηματοδότησης που δεν έχουν όλοι τους ίδιους κανόνες και την ίδια κρατική ενίσχυση. Κάποιοι λοιπόν δικαιούχοι προσπαθούν να συνδυάσουν ε, το Ταμείο Γιούνκερ με το πρόγραμμα ορίζοντας, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα τέλειων συνεργειών, αλλά νομίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να μας στείλει η Κομισιόν κάποιες σημειώσεις. Ε, αλλά η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν και θα πρέπει να έχουμε και άλλα κίνητρα για ολοκληρωμένη χρήση για την επόμενη περίοδο. Λοιπόν, τέλος, ε, πριν ε, το τέλος τα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως σας είπα, αυξήθηκαν από το 11% στο 44% χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι. Θεωρούν πως οι πλουσιότερες χώρε θα έπρεπε να έχουν κάποια υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν με τρόπο ανακυκλούμενο κάποια από αυτά τα κονδύλια, αλλά έτσι θα έχουμε απλά περισσότερους κανόνες. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τα κονδύλια αυτά και για τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις. Θα είναι έτσι για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα είναι πιο ελκυστικό. Επίσης, ε, οι μηχανισμοί δεν γνωρίζονται θα έλεγα αρκετά καλά, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Συνοψίζοντας, Νομίζω πως ε, κάναμε καλύτερη δουλειά το 2014-2020 για να ε, έχουμε προγράμματα αποτελεσματικά. Λειτουργήσαμε με καλό τρόπο, αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερος ακόμα. Υπάρχει λοιπόν ακόμα ε, η δυνατότητα όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα σύμφωνα με τα στοιχεία να αυξηθεί το ποσοστό εκείνο το οποίο βασίζεται στην απόδοση και να πάει μεγαλύτερο κομμάτι, όπως είπα, να είναι εξαρτώμενο από την απόδοση, λιγότερους περιορισμούς για χρηματοοικονομικά μέσα, να συνεχίσουμε τη θεματική εστίαση, να δοθούν κίνητρα για συνέργειες μέσω της εναρμόνισης ταμείων και της μείωσης των φραγμών μεταξύ διευθύνσεων και βέβαια όσον αφορά τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και να αξιολογήσουμε αν υπάρχει πρόσθεμενη αξία στους τρεις μηχανισμούς ε, παροχής αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να μπει νομίζω το ίδιο έργο και στον ορίζοντα 2020 και στο ε, Ταμείο Γιούνκερ και στα διαρθρωτικά ταμεία και να δούμε αν υπάρχει κάποια προσθεμένη αξία για να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί σε βάθος χρόνου. Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις από εμένα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος αγορητής, κύριος Χάιλ, Πίτερ Χάιλ, διευθυντής Αλτούς από την Ουγγαρία. Να υπενθυμίσω κάτι. Έχουμε όριο 10 λεπτών για τις παρεμβάσεις εκάστου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, ε, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ και εγώ από πλευρά μου που μπορώ να σα προσφωνήσω σήμερα. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρονικό όριο των 10 λεπτών που μου δώσατε. Το δικό μου επαγγελματικό σκηνικό ποιο είναι. Εργάστηκα για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία εδώ και πολλά χρόνια. Έχω αναλώσει δύο πλήρεις ε, προγραμματικές περιόδους με τα διαθροτικά ταμεία μεταξύ 2004 και 2013. Πρόσφατα εργάστηκα ως σύμβουλος και μάλιστα και σε ε, λοιπόν, ε, Οι γνώσεις μου αφορούν αυτό το επίπεδο και αυτά τα οποία θα αναφέρω ευελπιστώ ότι θα δείτε ότι σχετίζονται συνολικά σφαιρικά με τα θέματα του νέου κανονισμού. Σε σχέση με τους κανονισμούς αυτούς, άμα τους διαβάσετε, θα συμφωνήσετε πιθανότητα μαζί μου ότι υπάρχουν τρεις κυριότερες πτυχές όπου υπάρχουν ουσιοδός ε, νέες πρωτοβουλίες που προδιαγράφονται. Πρώτον, ο κανονισμός επικεντρώνεται στην επίτευξη των πρώτα και κύρια στο πλαίσιο της πολιτικής για την Ευρώπη του 2020, του ορίζοντα 2020. Ενδυναμώσαμε περιφερειακές προσεγγίσεις σε όλα τα περιφερειακά επίπεδα από τις μακροπεριφέρειες ε, και πολυσχηδώς σε όλα και πάλι θέτουμε το κέντρο βάρους στον καλύτερο συντονισμό των κονδυλίων των ταμείων και αποτελεσματικότερο, αποτελεσματικότερη διαχείριση. Φυσικά όσοι έχετε πείραση με όλα αυτά τα θέματα θα πείτε τίποτα από όλα αυτά δεν είναι απόλυτα καινοτόμο και καινούριο, καινοφανές και προερχόμενος από την Ουγγαρία δεν είναι τίποτα θεμελιωδώς καινοφανές από όλα αυτά. Θα μπορούσε κανείς να πει και για την περιφερειακή προσέγγιση ότι είχαμε τουλάχιστον κάποιες από τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές ήδη πριν από το 2014. Είχαμε ήδη εξειδικευμένα προγράμματα για περιφέρειες όπου γεωγραφικά μειονεκτήματα είχαν σωρευτεί ή είχαμε και γεωγραφικά μειονεκτήματα και σε σχέση και με το Λίντερ και το μέσο ανάπτυξης, το περιφερειακό μέσο ανάπτυξης και στην Ουγγαρία όχι μόνο είχαμε περιφερειακά προγράμματα αλλά και προγράμματα εξειδικευμένα για την αντιμετώπιση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να αναφερθούμε σε σχέση με τον ε, κανονισμό ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες λεπτομέρειες, ε, πολύ περισσότερη αρρωγή συνδρομή μπορεί να δοθεί ώστε να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση των κρατών μελών και για τις απαιτήσει όσον αφορά την χρηματοδότηση τρίτων σε σχέση με τον ε, συντονισμό και την διαχείριση Όλοι γνωρίζουμε ότι η απλούστευση ήταν ε, ένα μόνιμο διαρκές ε, αηφόρο στοιχείο. Έχουμε κάνει πιστεύω και πάλι σημαντικά βήματα εδώ προς αυτήν την κατεύθυνση. Η απλουστευμένη μορφή όσον αφορά την επιλογή κόστους ε, και τις διατάξεις για την χρήση ηλεκτρονικής διαχείρισης όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων που ευελπιστώ ότι θα καταστούν πραγματικότητα σε λίγα χρόνια, σε μικρό χρονικό διάστημα. Συνολικά Συνολικά δεν επινοήσαμε λοιπόν εκ νέου τον τροχό από το 2014 στο 2020, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία έχουν μετεξελιχθεί περαιτέρω σε συστηματική βάση. Εδώ υπάρχει εξειδίκευση μέσων και εργαλείων και όλα αυτά που έχουμε στην ε, οθόνη τώρα συνδέονται μεταξύ τους με το, την ε, επιθυμία να επιτευθεί ο στόχος, δηλαδή πρόσθετη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επικεντρωθούμε σε χειροπιαστά βελτιωμένα αποτελέσματα. Πώς όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν. Αν δούμε τις, ε, τα τρέχοντα προγράμματα όσον αφορά τη λειτουργία τους θα δείτε ότι σε πολλά μέρη, σε πολλά τμήματα έχουν αλλάξει και είναι και πάρα πολύ σύνθετα και περίπλοκα από την άλλη πλευρά. Επίσης σημειώνοντας ότι η κύρια ύπαρξη δεν είναι σε, έντυπο, σε έντυπη μορφή αλλά η ηλεκτρονικά πολύ καλά αν είσαστε εξειδικευμένοι ειδικό με υπολογιστές αλλά γιατί διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς όλα αυτά τα στοιχεία ηλεκτρονικής αποθήκευσης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του μη ολοκληρωμένου γάμου, του συνδυασμού, του προγραμματισμού και της υλοποίησης. Μέτρων δηλαδή που κάναμε πάντα, ε, διαχειριζόμαστε τα προγράμματά μας. Δεύτερον, η προσέγγιση η οποία επικεντρώνεται θεματολογικά σε προτεραιότητες επενδύσεων και σε συγκεκριμένους στόχους ή αποτελέσματα που πρέπει να δώσουν αυτά τα προγράμματα. Και τα δύο είναι αναγκαία ως συνιστώσεις. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι όπως ε, έγιναν αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μας αποθαρρύνουν στο να καταλάβουμε τι κάνουμε με αυτά τα προγράμματα και να δούμε πώς μπορούμε πιο εξειδικευμένα και πιο ε, εξειδικευμένα και ε, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια να δούμε τα, τα στοιχεία που αποθηκεύονται αποθηκεύονται στοιχεία τα οποία περιπλέκουν κάπως τη διαδικασία υλοποίησης γιατί αν θέλετε να μάθετε για τα αποτελέσματα απαιτείται ένα πολύ σύνθετο πλαίσιο στοιχείων αναφοράς και άντλησης. Υπάρχει εδώ ο κίνδυνος να υπερβούμε τα εσκαμένα και να καταχραστούμε αυτών των δυνατοτήτων και αυτό να αποβεί βάρος μας. Να υπενθυμίσω εδώ σε σχέση ε, με ε, εν παρενθέσει αυτό που έκανα ήταν είχα δώσει έδινα συμβουλές ε, στις ε, υποένταξη χώρες και χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων υπό το πρίσμα της περιφερικής ανάπτυξης είχαμε ήδη μια πολύ καλή προσέγγιση και κατανόηση με το σύνολο κανόνων και ρυθμίσεων ωστόσο για αυτά τα κράτη θα πρέπει να δούμε το περίπλοκο του χαρακτήρα και να μην αποτραπούν από το να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Αν προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα θα έλεγα ότι συνολικά υπάρχει σημαντική ευθυγράμμιση με την Ευρώπη 2020. Αν δούμε τι γίνεται με την Ουγγαρία, οι προτεραιότητες άλλαξαν σε τόσο σημαντικό βαθμό μεταξύ της περίοδου 2007-2014 που σχεδόν υπάρχει ο πειρασμός να πω ότι άλλαξαν περισσότερο από ότι άλλαξε η ίδια η Ουγγαρία ως χώρα. Δεύτερον, έχουμε μια λογική η οποία είναι κάθετη και σαφέστατη, είναι πιο αξιόπιστα και καλύτερα προπαρασκευασμένα τα προγράμματα πλέον. Αληθεύει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σε θέση πολύ αποτελεσματικά να διαπραγματευτεί με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή η Ευρώπη 2020 και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο είναι στοιχεία παρόντα σε όλα, σε όλες τις δράσεις και πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό. Από την άλλη πλευρά φυσικά υπήρχαν σημαντικότατες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τα κράτη-μέλη. Όλοι είχαν υποστεί αυτή την πίεση από την αλλαγή στοιχείων για τις επιδόσεις, ίσως ήταν τεχνικού χαρακτήρα θέματα, αλλά και για τους πραγματογνώμονές μας ήταν καινοφανή όλα αυτά. Και θα έλεγα ότι όλα αυτά καταδεικνύονται από το γεγονός ότι η προγραμματική διαδικασία καθυστέρησε κατά ένα έτος σε σχέση με σύγκριση για την περίοδο του 2007 όπου πάλι υπήρξε ε, μια επιβράδυνση. Την επόμενη φορά θα πρέπει να επιταχύνουμε το προγραμματισμό για να μην χάνουμε χρόνο και ευκαιρίες ε, ήδη από την έναρξη των προγραμμάτων. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα εδώ τώρα. Αφενός, όπως σας προανέφερα, πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια να απλουστεύσουμε περαιτέρω την προγραμματική φάση έχουμε περάσει σε ένα πολύ σύνθετο και περίπλοκο εγχείρημα προγραμματισμού. Καταδείξαμε ότι μπορεί να λειτουργήσει, δημιουργήσαμε προγράμματα με σημαντική στροφή προς τα χειροπιαστά βελτιωμένα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει να επεξηγηθούν και στους πολίτες πέρα από τις, ε, τα στοιχεία τα οποία μπορεί να παρουσιαστούν για τις ε, προσδοκίες μας όσον αφορά τα αποτελέσματα, μια πιο εύληπτη παρουσίαση. Και μετά μπορεί κανείς να υποσχεθεί επί παντός του επιστητού ό,τι επιθυμεί στους πολίτες σε σχέση με τις αναφορές. Και πράγματι στα προγράμματά μας η υλοποίηση χειροπιαστή είναι εκείνη που θα κάνει όλη τη διαφορά. Σε ένα από τα δημοσιεύματα σε σχέση με αυτή την έκθεση από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής διάβασα ότι τώρα είναι δουλειά πλέον των κρατών μελών να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα. Μάλιστα, αληθεύει αυτό. Αλλά υπάρχει εδώ το θέμα της συνδιαχείρισης, της επιμερισμένης διαχείρισης. Θα πρέπει επιτόπου να παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τεκτενόμενα. Υπάρχουν αρκετέ δυνατότητε και φορεί μέσω των οποίων μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και να διαπιστώσει αν υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσει ή όχι. Τρίτο σημείο, μια συνολική παρατήρηση, σφαιρική παρατήρηση που πιστεύω ότι πάει λίγο παραπέρα από τα όσα αναφέρονται γραπτά στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεπερνά αυτά τα οποία αναφέρονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Πρόσφατα, τουλάχιστον στην Ουγγαρία, τη χώρα μου, είχαμε αρκετά πώς να το πω, δυσάρεστες ε, συζητήσεις για το θέμα της ε, πολιτικής συνοχής και των στοιχείων της. Και ενώ όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα θα συμφωνούσαμε ότι έχει διτή αποστολή αφενός να δράσει ως ένα επενδυτικό όργανο και μέσο πανενοσιακά για το σύνολο της Ευρώπης, από την άλλη πλευρά είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο έκφρασης αλληλεγγύης. Κάποιοι όμως στη χώρα μου είπαν, ε, όλα αυτά είναι πράγματα που απορρέουν από το ότι είμαστε ένα νέο κράτο μέλο δεν είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένα. Είναι ούτω ή άλλω δικαίωμά μα να έχουμε αυτά τα κονδύλια στην ε, υπηρεσία μα. Όχι, νομίζω ότι πρέπει εδώ να καταστεί σαφέ ότι η πολιτική συνοχή είναι ένα μέσο αλληλεγγύη. Είναι ένα μέσο για την όλο και μεγαλύτερη ε, προσέγγιση και σύγκληση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια όλο και μεγαλύτερη και στενότερη ένωση. Και συζητώντα τα θέματα του 2020 να μην ξεχνάμε ότι η πολιτική συνοχή είναι μια από τις πιο σημαντικές απαντήσεις στα δυσάρεστα και πιεστικά ερωτήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αν κάποιος ε, δεν ε, δείχνει αλληλεγγύη, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον για την πολιτική συνοχή. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Επόμενη ε, ομιλήτρια θα αναφερθεί περισσότερο στις σχέσεις ε, πολιτικής συνοχής ε, και περιβάλλοντος. Είναι η κυρία Ιρέν Λούσιους. Ε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να μιλήσω ε, στα λεπτά τα οποία έχω στη διάθεσή μου να αναφερθώ, για να αναφερθώ στην περιβαλλοντική διάσταση της πολιτικής συνοχής με μια ιδιαίτερη εστίαση στις νέες χώρες. Γιατί είναι τόσο σημαντικά τα διαφορετικά ταμεία για το περιβάλλον. Πρώτον, γιατί υπάρχει το στρατηγικό ε, πλαίσιο για την δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης. Ε, πρέπει να σας πω ότι η Διεύθυνο που είναι εκπροσωπώ πριν από μερικά χρόνια ε, έκανε μία μελέτη σχετικά με την δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Επίσης, μέσω των, μέσω των πόρων αυτών, γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθεί ε, η αποδοτικότητα των πόρων και να κινηθούμε προς μια ε, οικονομία που θα καταναλώνει ε, λιγότερο άνθρωπο και θα έχει λιγότερες εκπομπές. Έχουμε 16 μελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι οι επενδύσεις έχουν γίνει πιο αποτελεσματικές και εστιασμένες. Επίσης ότι στηρίζεται ε, η πολιτιστική φυσική κρονομιά ε, και ότι τα νέα μέτρα συμβάλλουν ε, στην οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επίσης ότι η CLDD είναι ένα ισχυρό εργαλείο και ότι η προσέγγιση είναι καλά οργανωμένη αλλά θα πρέπει να οργανωθεί ακόμα περισσότερο γιατί το περιβάλλον δεν έχει ε, σύνορα και επομένως η συνεργασία θα πρέπει να είναι διαμεθοριακή και διαπεριφερειακή. Επίσης ότι χρειάζεται στήριξη από την Κομισιόν και ότι χρειάζεται απλουστευμένη πρόσβαση. Θα ήθελα λίγο να ε, ξαναδούμε ε, όλα αυτά τα μηνύματα. Ας αναφερθούμε πρώτα στην μεγαλύτερη εστίαση και στον καλύτερο προσανατολισμό τους στόχους δηλαδή. Η εμπειρία μας ε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δείκτες ας πούμε για τα προγράμματα Natura 2000 και οι στόχοι είναι ιδιαίτερα υπερβολικά ε, γενικευτικοί και επομένως δεν ε, προωθούν ε, για, στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Ε, μερικές φορές λείπουν κάποια δεδομένα όπως ας πούμε χάρτες, στοιχεία για την ενέργεια ε, και επομένως ε, δεν ε, γίνονται σωστές μετρήσεις. Ε, όσον αφορά τις αξιολογήσεις, ε, τις στρατηγικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και άλλου τέτοιου είδους ε, μελέτες, αυτές δεν είναι αρκετά σε βάθος ε, μπορούν να ε, ε, αποβούν εν τέλει αρνητικές προς το περιβάλλον γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος μέτρα, λανθασμένο σχεδιασμό. Έχουμε δει ας πούμε μια κακή, ένα κακό πρόγραμμα για την πλοήγηση στην Ρουμανία ή στην Ουγγαρία, ένα κακό πρόγραμμα όσον αφορά την προστασία από πλημμύρες αλλά βεβαίως ε, υπάρχουν και θετικές ε, εμπειρίες, παραδείγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μαθήματα για βελτίωση. Ε, όσον αφορά τώρα την βιο ποικιλότητα και το κλίμα και εδώ λείπουν κάποια στοιχεία. Το δεύτερο στοιχείο, μήνυμα ε, της ε, ε, έκθεσης αφορά το, την, εθνική, την, την περιβαλλοντική κληρονομιά, την κληρονομιά της φύσης. Πιστεύουμε ότι οι προτεραιότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην οδηγία για την προστασία προστασία των οικοσυστημάτων και των πουλιών. Επομένως, ε, χρειάζεται μεγαλύτερη εστίαση και εδώ. Επίσης, πιστεύουμε ότι η χρηματοδότηση της Natura 2000 θα πρέπει να γίνει πιο εξειδικευμένη ε, και ε, στόχο προσιλωμένη. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ορισμένοι, ορισμένες χρηματοδοτήσεις, ορισμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα δημιουργούν πρόβλημα στις περιοχές Natura 2000, υδρογεωλογικά, πούμε, με ε, υδρογεωλογικοί σχεδιασμοί όπως ανέφερα και προηγουμένως. Όσον αφορά την οικονομία χαμηλής χρήσης ε, άνθρακα για την ε, κεντρική Ευρώπη μονάχα ε, ε, χρησιμοποιούνται 6% για, από, τα, από τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής για προγράμματα διασφάλισης ενεργειακής αποδοτικότητας ή προγράμματα που εμπλέκουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι λυπηρό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι βλέπουμε ότι ακόμα ε, χρησιμοποιούνται πολλά χρήματα για υποδομές, δρόμους κλπ. Καθώς επίσης ε, και για, ε, και για ορυκτά καύσιμα. Όσον αφορά επίσης το ίδιο θέμα πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάποιες πολύ ευρύς, κάποιους πολύ ευρύς ορισμούς που εν τέλει δεν δημιουργούν κίνητρα για ε, ε, χρήση βιώσιμων τεχνολογιών. Ε, τα κριτήρια βιωσιμότητας, όπως είπα και προηγουμένως, λείπουν, π.χ. για την περίπτωση βιομάζας. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν καλά μέτρα όσον αφορά την χαμηλή χρήση άνθρακα και την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά στην ουσία αυτό αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ε, οι κλιματικοί στόχοι να ε, ε, είναι παρόντες σε κάθε είδους επένδυση, ας πούμε ακόμα και είναι μια επένδυση για τον τουρισμό. Τα CLLD και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές άραγε λειτουργούν. Επ' αυτού μπορώ να πω τα εξής πολύ συχνά βλέπουμε ότι η ικανότητα των εμπειρογνωμόνων ή η πραγματογνωμοσύνη συχνά είναι ανεπαρκή και επίσης ότι η επιλογή, η διαδικασία επιλογής των ε, projects δεν είναι αρκετά διαφανής, θα πρέπει να βελτιωθεί. Όταν μιλάμε τώρα για τις ε, ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ε, θα πρέπει να σας δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε ε, το διαμεθοριακό πρόγραμμα για τον ε, Δούναβη είναι της τάξης των 71 εκατομμυρίων αλλά μονάχα 27% αναφέρεται σε στοιχεία που άπτονται του περιβάλλοντος. Δηλαδή έχουμε καλά προγράμματα αλλά με μικρή χρηματοδότηση για το περιβάλλον. Στήριξη τώρα από πλευρά της Κομισιόν όντως χρειάζεται αυτή η ε, στήριξη. Συχνά διαπιστώνουμε ότι ε, δεν υπάρχει η δυνατότητα ε, αξιολόγησης των project ή δεν υπάρχει η απαραίτητη ικανότητα ή τεχνογνωσία εστίασης, κυρίως για προγράμματα βιοπικιλότητας και που σχετίζονται με το κλίμα. Ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για ανταλλαγές, ε, ανταλλαγή γνώσης, ε, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στοιχεία που θα αφορούν το περιβάλλον ή το κλίμα και που θα πρέπει οπωσδήποτε να κυκλοφορούν μεταξύ των χωρών. Χρειαζόμαστε άραγε απλουστευμένη πρόσβαση, η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν συνθήκες οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολες ε, όσον αφορά την πρόσβαση σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αναφέρομαι ας πούμε σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η προχρηματοδότηση. Ε, σε άλλες περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει και περιορισμένη πρόσβαση όπως ας πούμε ε, στην Ουγγαρία όπου μπορεί να επιλέξουμε με διοικήσει μονάχα των εθνικών πάρκων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΦΣΥ είναι ε, ιδιαίτερα γραφειοκρατική και δεν αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια για καλή υλοποίηση να κάνω και κάποιες ε, γενικότερες σκέψεις ε, σχετικά με τον πώς οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα. Ε, τώρα έχουν την δυνατότητα ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή Επιτήρησης Monitoring ε, Committee και μπορούν να παράσχουν συμβουλευτικές δραστηριότητες. Αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης μπορούν να παράσχουν μαζί με άλλες οργανώσεις πολιτών τεχνογνωσία. Σε εν λοιπόν οι συστάσεις μας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι επενδύσεις να γίνουν πιο αποτελεσματικές, να έχουν μεγαλύτερη αστίαση, ε, ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η λογική των παρεμβάσεων ε, και επομένως να έχουν καλύτερη στοχοπροσύλωση και ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, ε, τα κίνητρα να είναι σωστά έτσι ώστε να επιλέγονται σωστά και οι στόχοι. Επίσης, τα, οι δείκτες αποτελέσματος θα πρέπει να τυποποιηθούν καλύτερα, ας πούμε, για την εξοικονόμηση ενέργειας και βεβαίως σε επίπεδο προγράμματος θα πρέπει να διατίθενται δημόσια οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Είναι καλό να διατηρήσουμε την εστίαση στο Natura 2000 αλλά πιστεύουμε ότι όσον αφορά εξειδικευμένες ανάγκες ε, θα πρέπει να έχουμε και πιο εξειδικευμένη προσέγγιση. Θα πρέπει επίσης τα CLD να ε, λειτουργήσουν ε, με την συμπερίληψη και πραγματογνωμόνων και επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί οπωσδήποτε η διαφάνεια των διαδικασιών. Θα πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι σε διαμεθοριακά προγράμματα. Ε, επίσης να μην δίνονται πλέον επιδοτήσεις ε, για ορυκτά καύσιμα ή τέτοιες σχετικές τεχνολογίες, ούτε ε, για κλασικά προγράμματα υποδομής, δημιουργία δρόμων κλπ που μειώνουν το φυσικό κεφάλαιο. Επίσης χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη από την Κομισιόν να ε, υπάρχει επομένως ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά ε, το κλίμα, όσον αφορά την ε, βιοδιαθεσιμότητα και να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση και εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τέλος πιο απλουστευμένη προσέγγιση για όλους τους φορείς και ιδίως για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκόργ, ε, Γκορζελάκ, δεν ξέρω αν το πρόφερα καλά. Ε, ο κύριος Γκορζελάκ ε, είναι, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είναι πραγματική πρόκληση να προσφωνεί κανείς ένα τόσο απαιτητικό ακροατήριο. Θα κάνω λόγο για αυτό που θεωρώ ότι τεκταίνεται στην κεντροανατολική Ευρώπη, στα νέα κράτη-μέλη και πώς η πολιτική συνοχή μπορεί να συνεισφέρει από πλευρά τη συμπεριλαμβανομένων και των ευκαιριών ε, για να είναι οι χώρες αυτές πιο ανταγωνιστικές σε μια παγκοσμιοποιημένη ανοιχτή οικονομία. Πρώτα απ' όλα να δούμε αυτό το γράφημα που δείχνει ότι συνολικά μετά από το 1990 ήταν επιτυχής αυτές οι χώρες. Σημείωσαν αύξηση, πολλές διπλασίασαν το ΑΕΠ τους και βλέπουμε ότι υπήρξε αυτή η μετατροπή, η μεταμόρφωση. Η ουσία όμως αυτή είναι. Αν δείτε μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη επιτυχία στην κεντροανατολική Ευρώπη βρίσκεται. Διότι ακόμα και η χειρότερη κεντροανατολικοευρωπαϊκή χώρα είναι καλύτερη από τις επιδόσεις των κεντροδυτικών ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα μετά το 2004. Και κάποιες χώρες όπως η Σλοβακία για παράδειγμα, η Πολωνία, μπόρεσαν να, να ξεκινήσουν ακόμα περισσότερο και να πάνε ακόμα πιο μακριά με το ποσοστό ανάπτυξής τους σε σχέση για παράδειγμα με το ποσοστό ανάπτυξης τη Σουηδία ή της Αυστρίας ή των δυτικών χωρών της ευρωπαϊκή Ένωσης. Αυτό όμω μπορεί να διατηρηθεί ε, για πάντα αυτό είναι ένα ερώτημα που διατυπώσαμε στη μελέτη μας. Ε, είχαμε 27 ε, παρατηρήσεις ε, που έγιναν, μελέτες που έγιναν. Η απάντηση είναι όχι. Είναι αρνητική. Όχι. Δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Υπάρχουν προκλήσεις οι οποίες ε, αντιμετωπίστηκαν, βρέθηκαν μπροστά σε αυτές τις χώρες και έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Πρώτον, η επιτυχία βασίστηκε σε εξωτερικούς πόρους. Ε, ε, τα περισσότερα κονδύλια ήρθαν εκ των έξω. Η καινοτομία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και με την εξαίρεση της Σλοβενίας βρισκόμαστε στο κάτω τμήμα της καινοτομία ε, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξωτερικές πηγές ε, ε, ανταγωνιστικότητας στις οποίες βασίστηκε η επιτυχία μας είναι χαμηλή μισθή χαμηλό κόστος παραγωγής σε σχέση με τους ε, ανταγωνιστές μας ε, που βρίσκονται δίπλα μας, για παράδειγμα την Ουκρανία ή και την Απαρατολική δημογραφικές προκλήσεις ε, με πολύ χαμηλό ποσοστό φυσικής ανάπτυξης και υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος συνταξιοδότησης. Δεν είμαστε εμείς μοναδικοί με αυτές τις ιδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Βρισκόμαστε όμως στην άκρη, στα και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ε, υπάρχουν πολλά θέματα για το περιβάλλον και δεν θέτουμε ιδιαίτερα κέντρο βάρους ε, σε αυτή τη συνιστόσα της ανάπτυξης. Ε, η παγίδα του μέσου εισοδήματο, που είναι η παγίδα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαφύγει κανείς από αυτήν σε σχέση για παράδειγμα με τα 15.000 δολάρια ανακάτοικο. Για θέλουμε να βγούμε έξω από αυτήν την παγίδα για την καινοτομία και να βασίσουμε την ανάπτυξή μας σε ένα διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης είναι μεγάλη πρόκληση και την έχουμε ενώπιόν μας. Τώρα σε ποιο βαθμό οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης που έχουν βέβαια συνταχθεί στα χαρτιά, αλλά αυτά τα θέματα κατά πόσον υλοποιούνται στις στρατηγικές μας και στα προγράμματά μας ε, στην εφαρμογή των πολιτικών συνοχής. Πρώτον, υπερβολική, ε, ε, υπερβολικό κέντρο βάρους στις υποδομές και πολύ λίγο κέντρο βάρους θέτουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να δούμε ότι οι, οι ήπιες υποδομές, θεσμικά όργανα, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, το κοινωνικό κεφάλαιο του ανθρώπινου δυναμικού, αυτά αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Επικεντρωνόμαστε ή παρεκκλίνουμε όσον αφορά την χρήση των διαθωτικών ταμείων και των κονδυλίων. Έχουμε κάποια παραδείγματα σε σχέση με νοτιοευρωπαϊκά κράτη τα οποία βρέθηκαν στην παγίδα της χαμηλής αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας αυτά τα κονδύλια. Κατά κάποιο βαθμό ακολουθούμε και εμείς αυτή την τάση. Διότι υπάρχει μια αύξουσα τάση ότι όλοι λέει πρέπει να υποφεληθούν. Θα επανέλθω σε αυτό το σημείο υστερότερα και θα τοποθετηθώ επ' αυτού. Στρατηγικές όσον αφορά τώρα την έρευνα και την ανάπτυξη με βάση τις έδρες στα κράτη-μέλη και πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτή η πολιτική έρευνας και ανάπτυξης ε, θα ακολουθηθεί. Διαφορετικά αν δεν ε, συγκλίνουμε τότε θα αυξηθούν οι διαφορές. Πρέπει εδώ να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια συνέχεια θα δώσουμε στην πολιτική έρευνας και ανάπτυξης. Σπουδαιότητα της τελευταίας γραμμής εδώ σε αυτό το γράφημα. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι αλληλεξαρτήσεις και οι κειμεν... κειμενόμενες σχέσεις μεταξύ ε, των χωρών χωρών μας όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι άγνωστα αυτά τα στοιχεία όσον αφορά και την κοινή αγροτική πολιτική. Θα επανέλθω σε αυτό το σημείο υστερότερα μετά περιβάλλον. Κάποιες χώρες όπως η δική μου χώρα έχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις να ακολουθήσουν την οδό της αποανθρακοποίησης, της μείωσης των εκπομ της χρήσης άνθρακα και των εκπομπών και επιβάρυνσης του ατμοσφαιρικού αέρα με άνθρακα. Ε, αυτό όμως δεν είναι μόνο περίπτωση, η περίπτωση της Πολωνίας. Υπάρχουν και άλλες χώρες ε, που έχουν αυτές τις επιφυλάξεις. Ε, εισάγουμε πολλά παλαιά οχήματα αντί να αγοράσουμε καινούρια οχήματα και αυτό είναι πρόβλημα το οποίο επιβαρύνει ακόμα περαιτέρω το περιβάλλον, τον ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης έχουμε πολλά παραδείγματα υπερεπένδυσης ε, όσον αφορά την ε, περιβαλλοντική συνιστόσα. Για παράδειγμα όσον αφορά τα απόβλητα ή τα λύματα. Και εδώ πρέπει να δούμε σε σχέση με τις δομές ε, που μπορούν να δημιουργηθούν με τα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων να μην επιβαρύνουν ή παραλύσουν δήμους και κοινότητες που δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια πορεία ανάπτυξης ε, με τέτοια επιβάρηση για την ε, απασχόληση επιβράδυνση απασχόλησης και η απασχόληση των νέων επιβραδύνεται περισσότερο από τις άλλες χώρες βρισκόμαστε χαμηλότερα, σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι ε, όσον αφορά την πολιτική απασχόληση σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε επαρκώς αναπτύξει την διαβίου κατάρτιση και εκπαίδευση που θα έπρεπε να είναι ένας από τους στόχους της πολιτικής συνοχής και που θα έπρεπε να διευρυνθεί μέσω αυτής ε, ο στόχος. Και μετά σε κάποιες χώρες υπάρχει εθνοτικό πρόβλημα πολύ θα έλεγα πολυδιάστατο πρόβλημα μειονεξιών και ε, αρνητικής θέσης στην οποία βρίσκονται μειονότητες όπως για παράδειγμα οι Αθήγανοι, ο πληθυσμός Ρωμά, οι Τσιγκάνοι. Δεν έχει επιληθεί αυτό το πρόβλημα, διευρύνεται και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο, οξύνεται περισσότερο με το φαινόμενο της μετανάστευσης θεσμική σύγκληση. Βρήκαμε στην έρευνά μας ότι τα προβλήματα σε σχέση με την θεσμική σύγκληση ε, μετά το 2003 ε, έχουν, ε, έχουν πλέον παγιωθεί. Η πρόοδος είναι χαμηλότερου επίπεδου από ό,τι πριν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την ομάδα έρευνας θεσμικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα εξάρτησης και άλλη εξάρτησης που δεν αναπτύξαμε μόνο εμείς διότι αφορά όλα τα διεθνή προγράμματα σε σχέση με την χορήγηση αρρωγής. Αυτό το όμως το φαινόμενο εξάρτησης από εξωτερική αρρωγή όπως σημειώνεται και στην Πορτογαλία και τώρα διαπιστώνεται και στην κεντροανατολική Ευρώπη διότι η Πορτογαλία είναι η περισσότερο εξαρτημένη χώρα από κονδύλια, ευρωπαϊκά κονδύλια όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις οι επόμενες χώρες στην κλίμακα μετά την χαμηλότερη την Πορτογαλία είναι κέντρο ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά επηρεάζουν τις ικανότητές μας να μπορέσουμε να πάρουμε τα, το μέλλον μας, ε, το πεπρωμένο μας στα χέρια μας και να α, ε, μην εξαρτώμαστε από άλλους. Είναι ένα θέμα διαρθρωτικό και ένας ψυχολογικός παράγοντας κινδύνου. Είναι ένας α, ε, παράγοντας α, εξάρτησης κοινωνικής ψυχολογίας. Ίσως οι κοινωνικοί ψυχολόγοι θα μπορούσαν να επεκταθούν περισσότερο. Υπάρχουν όμως εδώ τάσεις πολιτικών που ακολουθούνται και καμιά φορά θεωρεί κανείς, μπορεί να θεωρεί κανείς ότι είναι εύκολα λεφτά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη που ήμουν τόσο επικριτικός, αλλά αυτή είναι η, είναι, αυτή είναι η αδυναμία μου. Πάντα πρέπει να είμαστε ευθύ και ειλικρινεί και να αναγνωρίζουμε ότι υφίστανται προβλήματα στην πολιτική, στην ε, γεωργική πολιτική. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ποια είναι τα προβλήματα και μετά να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το νόημα αυτής της παρουσίασης πολιτισμού σήμερα. Και αυτό όχι μόνο σε σχέση με συμφωνίε εταιρική σχέση όσον αφορά τι δομέ στι χώρε κεντροανατολικοευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει κάποια περιφερειακή σύγκληση. Ωστόσο όμω υπάρχει και μια αστικοποίηση, επικέντρωση στα αστικά κέντρα. Ο μεγαλύτερο παράγοντα δημιουργία ανισοτήτων για τα Ευρωπαϊκά κράτη. Α, χτύπησε ο συναγερμό. Να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω σιγά σιγά για την, ε, για την ε, συνοχή και όσον αφορά την ψυχολογική προσέγγιση μας ε, για την πολιτική συνοχή. Έχουμε τώρα ένα πρόγραμμα και ο Μπάτλερ που ήταν αρμόδιος για αυτή τη συνιστόσα θα εξετάσουμε μαζί ποιες είναι οι τάσεις και οι προσεγγίσεις, η αντιμετώπιση των κοινωνιών των κρατών μελών στην πολιτική συνοχή στο σύνολο των 28 κρατών μελών. Ίσως μετά από 1,5 χρόνο ακριβώς θα έχουμε πιο αξιόπιστα στοιχεία και συμπεράσματα στα οποία να βασιστούμε. Αξιολόγηση <clears throat> λιγότερο ε, τυπικού χαρακτήρα και περισσότερο ουσιώδης. Το λέγαμε αυτό εδώ και χρόνια ότι πρέπει να ενταχθεί η αξιολόγηση ενεργά στις ε, δράσεις μας και να μην κατακαιρματιστούμε και εξετάζουμε το Ταμείο την πολιτική συνοχή ξεχωριστά κατακαιρματισμένα με τις διάφορες διευθύνσεις πρέπει να πάμε κάτω επί και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις όλων των επεμβάσεων και ε, της παρεμβατικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι τα αποτελέσματά τους και υπάρχει μια θετική μεθοδολογική προσέγγιση επιστημονικά για να το κάνουμε αυτό. Όταν όμως έχουμε συσσωρευτικές ε, επιπτώσεις ε, ε, από πλευράς Υπουργείων ή πολιτικών έχουμε και τις ίδιες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να τις υπερβούμε, να τις ξεπεράσουμε. Η πολιτική συνοχή δεν πρέπει να χάσει, να απεμπολίσει την στρατηγική της προοπτική και να είναι ένας μηχανισμός και ε, να μην κινηθεί προς ε, ένα μηχανισμό ε, συγκυριακής αντιμετώπισης προβλημάτων και προκλήσεων. Εδώ πρέπει να είμαστε πιο ουσιώδεις και οι κεντροανατολικοευρωπαϊκές χώρες πρέπει επίσης να επωφεληθούν από δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την Connecting Europe, Europe Facility, τον μηχανισμό διασύνδεσης των ε, ε, χωρών της Ευρώπης μεταξύ τους, είτε στις μεταφορές, είτε στην ενέργεια, είτε αλλού. Πάντα όμως θα υπάρξουν και κάποιες αντιρρήσεις ή ενστάσεις από πλευράς κρατών που βρίσκονται ίσως στο περιθώριο γεωγραφικά βρίσκονται στις παρυφές ή εσχατιές με χαμηλότερο ποσοστό δυναμικού για την έρευνα και την ολοκλήρωση και ίσως αυτό μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα υποφελές και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό και να συμπεριληφθούν και αυτές οι χώρες. Η στρατηγική στόχη της Ευρώπης 2020 δεν θα έπρεπε μηχανιστικά, με μηχανικό τρόπο, ε, με τη φροσούρτη να υλοποιούνται σε σχέση με τις ε, προτεραιότητες, 11 προτεραιότητες σε όλες τις περιφέρειες όταν έχουμε επαφές και συζητούμε αυτά τα θέματα η ευφυής εξειδίκευση είναι ένα σημαντικό θέμα. Χρειάζεται όμως και ευφυής μη εξειδίκευση, ευφυής αντιμετώπιση δηλαδή των προβλημάτων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Να μην δούμε δηλαδή ε, την, ε, το ένα να προηγείται του άλλου. Πρέπει να υπάρχει ένα είδος, ε, ας το πω έτσι, πιο αποτελεσματικής και ορθολογικής προσέγγισης στα προγράμματα αυτά για τη συνοχή και την ανάπτυξη των χωρών μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές ήταν οι παρουσιάσεις ε, των ε, προσκεκλημένων μας και σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι ήταν ε, χρήσιμες και ενδιαφέρουσες. Τώρα θα δώσουμε τον λόγο στους βουλευτές. Κύριε Φανίστελ Ρόι, θα πάρετε τον λόγο στο τέλος. Εντάξει, σας πειράζει. Θα ήθελα, η πρώτη μου ερώτηση είναι αν θα λάβουμε τυπωμένες τις παρουσιάσεις. Έχουν ήδη μοιραστεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, λέει η Πρόεδρος. Α, θα μοιραστούν. Θα μοιραστούν μετά το τέλος της συνεδρίασης, με συγχωρείτε. Ωραία. Ε, φαντάστηκα ότι τι είχαν μοιράσει. Ε, αυτή δεν είναι ερώτηση, φαντάζομαι. Δεν μετράει στις ερωτήσεις μου. Εντάξει. Όχι, όχι, δεν, ε, δεν σας αποκλείει κανείς από τις ερωτήσεις. Ε, είναι σημαντικός ο ρόλος σας να κάνετε τελευταίος τις ερωτήσεις και θα λάβετε πρώτος απαντήσεις. Λοιπόν, κύριε Φανίστε Λοιπόν, ερωτήσεις, άρα όχι συμπεράσματα. Έμαθα αρκετά πράγματα λοιπόν για την ε, αποειδίκευση για την κοινωνική πτυχή της πολιτικής συνοχής, για την παγίδα του μέσου εισοδήματος. Ε, πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε και σας ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις λοιπόν. Λοιπόν, κανείς δεν μίλησε για την κοινή διαχείριση. Επιμερισμένη διαχείριση. Επιμερισμένη διαχείριση. Τι είναι. Να μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό. γιατί είπατε πως θέλετε κάποια προγράμματα τα οποία θα κατευθύνονται από τις Βρυξέλλες για λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό προς όλους τους ε, ομιλητές. Μετά για την ε, εδαφική συνεργασία. Το ακούσαμε μάλιστα στην ε, παρουσίαση για τον Δούναβη. Ενδιαφέρον αυτό. Γιατί εάν είναι πολύ ευρύτερη η ζώνη είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς συγκεκριμένος για τα αποτελέσματα της παρέμβασή του. Οπότε ίσως μάθουμε κάτι για την εδαφική συνεργασία και την εδαφική κλίμακα. Και η τρίτη μου ερώτηση επίσης αφορά αυτή την συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Ε, ξεκίνησε αυτή η περίοδος. Είχαμε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που προσθέθηκε στον κανονισμό και λέμε τι μπορούν να κάνουν οι περιφέρειες για να συνεργαστούν, για να ξοδευτεί ένα τμήμα των κονδυλίων σε έξυπνη εξειδίκευση και συνεργασία κτλ. Και δεν ε, υιοθετήθηκαν αυτά δεν ασχολήθηκε κανείς. Ε, και τέλος, για τα επίπεδα. Ο Ολλανδός εκπρόσωπος είπε ότι ξοδεύουν περισσότερα παραδείγματος χάρη σε κάποιους στόχους όπως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επειδή ήταν καλά διαρθρωμένοι. Δηλαδή στην Ολλανδία η το κεντρικό κράτος διαχειρίζεται το ταμεία και εσείς είστε στο περιφερειακό επίπεδο. Πώς το διαχειρίζεστε αυτό. Σας στέλνουν λεφτά στην δική σας την περιφέρεια. Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις που είχα εγώ. Ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι. Έχετε κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Έχω αρκετέ ερωτήσεις, αλλά να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τα πράγματα. Βλέπω το χρονοδιάγραμμα λέει ότι μέχρι τις 6 και 15 ε, θα είναι οι ερωτήσεις. Δηλαδή έχουμε μισή ώρα ερωτήσεων. Δεν θέλω να πάρω το χρόνο των ε, μελών της Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να αναφέρω τρία πράγματα τα οποία προέκυψαν και τα οποία ίσως ε, οι πανελίστες μπορούν να συζητήσουν, να αναλύσουν περισσότερο. Έχουμε κανονισμούς, ε, κοινέ ε, ε, διατάξεις, οι οποίες δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες. Νομίζω ότι ο κύριος Ράκ ανέφερε αυτή την ασάφεια. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, οι πανελίστες θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος κατά αυτή την έννοια από τώρα δηλαδή και μέχρι το τέλος της προγραμματικής περίοδου ε, υπάρχουν κάποιες φάσεις ε, τις οποίες ε, θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε αν προκύψουν κάποια κενά εγκαίρως να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν κάποιες ερεσιμότητες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να μην τις θεωρήσει η Κομισιόν ικανό τόπο για ενδεχόμενες ανακλήσεις ή αναιρέσεις. Ίσως κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα ε, ξαναδούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε εύκολα στη φάση της υλοποίησης των προγραμμάτων. Τέλος, θα ήθελα να κάνω και μία γενικότερη ας πούμε ερώτηση. Ε, ο τελευταίος ομιλητής μίλησε για συνοχή, ο πρώτος μίλησε ε, για επενδύσεις κλπ. Γιατί πράγμα μιλάμε όταν αναφερόμαστε στην συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων. Τι ακριβώς περιγράφει αυτό. Ναι, έχουμε όμως και το δεύτερο ομιλητή, ο οποίος είπε ότι μιλάμε για την πολιτική επενδύσεων και αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με ερωτήσεις από τον κύριο Νίλσεν. Παρακαλώ, κύριε Νίλσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά, πολλά θα μπορούσε κανείς να πει. Και εκ μέρους της ε, σουηδικής ε, πείρας ή εμπειρίας ήταν ενδιαφέροντα να ακούσει κανείς όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ ήμουν δήμαρχος ε, στην προηγούμενη ζωή μου όμως ε, σε σχέση με την περιφερική ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του 90 στη δική μου περιοχή όταν σήμερα αναφέρεται ότι χρειάζονται απλουστευμένα προγράμματα για αυτό το έργο. Εγώ προσωπικά έκανα, είχα την εμπειρία ότι πολύ συχνά πολλά πράγματα θα έπρεπε να απλουστευτούν και να γίνουν απλούστερα. Δεν θέλουν όμως να καινοτομήσουν. Δηλαδή αναφέρθηκε, αναφέρεται εγώ έκανα αυτή την εμπειρία. Όσο περισσότερο εμπλέκεται σε αυτά τα προγράμματα κανείς, τόσο περισσότερο το βλέπει. Τόσο περισσότερο στο τοπικό, περιφερειακό επίπεδο πρέπει να τα βλέπουμε. Όχι μόνο σε σχέση με τις εθνικές αρχές και τους εμπλεκόμενους, αλλά και την οικονομία μας. Αλλά η υλοποίηση στο τέλος τέλος είναι πολύ καλύτερη, γιατί επειδή όλοι εμπλέκονται και συμμετέχουν και τραβούν το σκηνή Προ προς την ίδια κατεύθυνση και γι' αυτό φοβάμαι καμιά φορά όταν ακούω να απλουστευτούν λέει όλα ισοπεδωτικά μπορεί να γίνει αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να δημιουργήσει ίσως και προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Μαθητής παρακαλώ έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική παρουσίασή σας ε, ενός λέει κυρία Μαλέτιτς. Παρατηρούμε πολλές τις δυσκολίες και εμπόδια κόμματα στην πολιτική συνοχή ε, να ε, σημειώνονται. Αναφέρθηκε η μελέτη που καταδεικνύει ότι στην νοτιοανατολική Ευρώπη υπάρχουν ακόμα χαμηλότερα θεσμικά δυναμικά σε σχέση με την προενταξιακή περίοδο ε, σε χώρες και αναφέρατε στην παρουσίασή σας ότι υπήρχαν δυσκολίες ε, για την επικέντρωση σε χειροπιαστά αποτελέσματα στην πρακτική εφαρμογή και ότι είναι πολύ σύνθετος και περίπλοκος ο χαρακτήρας αυτών των ε, προγραμμάτων και ότι είναι πολύ δύσκολο με κάποια ε, στοιχεία και μόνο να γίνουν όλα αυτά κατανοητά και να είναι εύληπτα. Παρατηρώντας όλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι με κάποια προοπτική όταν ε, ε, συρρυκνώνεται και όταν χώρες δεν έχουν την ταχύτητα, την όθηση να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, μένουν πίσω και επιβραδύνουν. Για την περίοδο 2014-2020 τα προγράμματα με βάση το... Ε, τα, προγράμματα με βάση τον προϋπολογισμό με την επικέντρωση σε χειροπιαστά αποτελέσματα και πολλά άλλα που αναφέρθηκαν ουσιαστικά στα κράτη-μέλη έχουμε διαφορετικές μεθοδολογίες που ακολουθούνται με τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του εθνικού προγραμματισμού εκάστοτε, του εθνικού προϋπολογισμού όπως προγραμματίζεται. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος, μια, ένας τρόπος ε, προγραμματισμού και προπαρασκευής και υπάρχει δυσκολία να παρακολουθήσουν την πολιτική συνοχής ε, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και προγραμματίζεται. Ιδιαίτερα σε σχέση με την πολιτική συνοχής όταν έχουμε την σημαντική αρχή της σορευτικότητας ή προσθετικότητας και πρέπει να υπάρχει και συγχρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς με κονδύλια από τα κράτη-μέλη, πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν. Ε, είτε στο εθνικό επίπεδο, είτε στην, ε, στον προγραμματισμό όσον αφορά τον ε, προϋπολογισμό από, από ευρωπαϊκής πλευράς. Αν δεν υπάρχει η επαρκής χρηματοδότηση, οι επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς καθιστούν δύσκολο το να παρακολουθήσουν τα κράτη το επίπεδο συνοχής ε, που είναι ευκταίο. Θα έπρεπε από κοινού λοιπόν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απασχοληθούν. Ξέρω ε, δράτε σε πάρα πολλά κράτη-μέλη και ενεργοποιήστε, όμως θα πρέπει αυτό να το δείτε του σύνεγγυς σε αυτή τη διάσταση που σας παρουσίασα. Και εσείς κύριε Γκόζελάκα αναφέρατε την εξάρτηση από την εξωτερική βοήθεια, aid dependence. Είδα πρακτικά ότι πολλοί επιχειρηματίες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Ανέφεραν ότι είναι τόσο περίπλοκοι και σύνθετοι οι κανόνες και είναι τόσο μεγάλη επιβάρυνση για την παρακολούθηση, και τις επεξηγήσεις υλοποίησης ε, με τους όρους που πρέπει να ακολουθηθούν αυτών των κονδυλίων δεν είναι καθόλου εύκολο λοιπόν να αποδεχτούν και να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια και λένε καλύτερα όχι και βασίζονται σε σχέση με τις ε, κρατικές ε, ενισχύσεις και υπάρχει και χαμηλό ποσοστό ακόμα και 5% και λόγω του γεγονότος ότι χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια Βασιλεία τίθεται και το θέμα των επιτοκίων και μια και υπολογίζουν τα πάντα ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται στο μείον και αναζητούν χαμηλότερα επιτόκια χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση την οποία επομίζονται λόγω της περίπλοκης υλοποίησης και εφαρμογής των κανονισμών και κανόνων του ευρωπαϊκού επίπεδου. Δεν είμαι βέβαια απόλυτα ότι δημιουργείται η ίδια λοιπόν εξάρτηση σε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι πραγματικά η σωστή χρονική στιγμή να τα συζητήσουμε για το πρόγραμμα του 2014-2020 που έχει ξεκινήσει. Μπορούμε τώρα να παρέμβουμε και να το επηρεάσουμε. Ας κάνω κάποιες προτάσεις και δια ερωτήσεις ταυτόχρονα που θα ήθελα να διατυπώσω. Επιτρέψτε μου να θέσω τα εξής ερωτήματα. Κάναμε σε μεγάλο βαθμό λόγο για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σαν να επρόκειτο αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια να ε, υπήρχε για αυτά μια συγκεκριμένη απορροφητικότητα Πιστεύω ότι αυτή η τάση υφίσταται στα κράτη-μέλη και πρέπει να διασφαλίσουμε από πλευράς μας ότι η ιδιοκτησία εντός εισαγωγικών, η κυριότητα των κονδυλίων, διότι αν αυτά είναι στην κυριότητα του προϋπολογισμού πρέπει, υπάρχει η φιλοδοξία να ε, διασφαλιστούν και να σε εισαγωγικά εξασφαλιστούν. Πρέπει να προαχθεί η ε, τάση αυτή. Μέχρι ότου όμως διασφαλιστούν ή εξασφαλιστούν αυτά τα κονδύλια αφαιρούνται από τους Δήμους και κοινότητες και χρησιμοποιούνται αλλού. Δεν υπάρχουν δηλαδή κίνητρα για την ε, διασφάλιση, εξασφάλιση αυτών των κονδυλίων. Και στο τέλος έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και τα οποία παρατηρούμε στα κράτη-μέλη για τη διαφορετική διαχείριση κονδυλίων. Κάποια κράτη έχουν κεντροποιημένη μορφή διαχείρισης, η Λιθουανία και άλλα κράτη. Κάποια άλλα κράτη έχουν μια πιο χαλαρή μορφή ή μη αποκεντρωμένη και άλλες χώρες, η τρίτη κατηγορία, είναι χώρες που έχουν προχωρήσει στην αποκέντρωση και εκεί βλέπουμε τα καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ αυτών. Κάνω λόγο δηλαδή για τα τελικά χειροπιαστά, ανάγλυφα αποτελέσματα, διότι οι επιδόσεις αυτών των προγραμμάτων, η ικανοποίηση των πολιτών και μάλιστα τα αποτελέσματα προς όφελος των ε, περιφερειών, Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι κοινότητες δεν εμπλέκονται έγκαιρα όπως θα έπρεπε. Πρέπει να συμφωνήσω με αυτή την πτυχή πρέπει να συμμετέχουν να ευθύ εξ αρχή στον προγραμματισμό και πρέπει να διασφαλίσουν τα μέγιστα ωφέλη. Ας αναφέρω το πρόγραμμα Leader για παράδειγμα ως προς αυτό. Υποδιαιρείται σαφώς και ίσως το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για την πολιτική συνοχή. Να κατανείμουμε 50% σε σχέση με τις κοινότητες και τους δήμους, 20% από επιχειρήσει, 30% ε, ή 50% από δηλαδή συνολικά 70% να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτά ποσοστοποιούνται, καθορίζονται για να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Στην πολιτική συνοχή όμως υπάρχει υπερβολικά μεγάλη διακριτική ευχέρεια, περιθώριο των κρατών μελών να λαμβάνουν αυτόνομα διαφορετικές αποφάσεις. Και έτσι αυτό στις ξεχωριστές φάσεις δημιουργεί προβλήματα. Είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και η διαφάνεια αυτή το ανοιχτός χαρακτήρας, η συνεργασία διατομεακά μεταξύ των εμπλεκόμενων θα διασφαλίζει αυτή την διαφάνεια που πάντα είναι επιθυμητός ευκταίος στόχος για μας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις αναφέρθηκε ότι επενδύουμε υπερβολικά πολλά σε χθεσινά σχέδια ή σε κάποια ε, προγράμματα και σχέδια με ε, προηγούμενο, ε, προηγούμενο παλαιότερο προφίλ Πρέπει όμως καινοτόμα, καινοφανή προγράμματα και σχέδια να, να, να προαχθούν όπως για τα ανανεώσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καινοτομία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Για παράδειγμα τώρα, σήμερα η Γαλλία έλαβε μία απόφαση πρόσφατα για ένα ελάχιστο μισθό ο οποίος ε, θα πρέπει να ε, λειτουργεί για τους μεταφορείς ε, μεταξύ των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος ε, έχει όμως ε, διαφορετικούς όρους, διαφορετική φορολογία, διαφορετικά εισοδή, ύψος, διαφορετικό ύψος εισοδήματος, ε, τελών και η ανταγωνιστικότητα είναι διαφορετική και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φανίστερβο. Ναι. Θα είμαι σύντομος για να υπάρχει και χρόνος να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Κοιτάξτε θα περιοριστώ σε μία ερώτηση, γιατί βεβαίως θα πρέπει η ανακοίνωση να αναφέρεται και στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, γιατί αναφέρθηκε η Κομισιόν στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Θεωρείτε ότι υιοθετήθηκε αυτή και πώς έγινε αυτό στην πράξη, γιατί δεν βλέπω κάτι στην ανακοίνωσή σας, κάποια ανάλυση της διαδικασίας. Δεν ξέρω, θα μπορούσατε να μας πείτε τις απόψεις σας για το θέμα. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Φαντούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για, την παρουσίαση που, για τις παρουσιάσεις που έγιναν εδώ πέρα. Θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, βεβαίως, Η έκθεση του άρθρου 16 είναι απλά το τι συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ έχουμε επιπλέον εξελίξεις και βλέπουμε πώς εξελίχθηκε ο κανονισμός και είδαμε κάποιες δυσκολίες με την ερεσιμότητα εξ άντε. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα, το λαμβάνουμε υπόψη. Και βεβαίως και για τις συζητήσεις μετά το 2020. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη. Από την παρουσίαση του κυρίου Φανεράκ συγκρατώ ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη έμφαση για τον συνδυασμό του ΕΦΣΥ και του ΕΣΥΦ για να υπάρξουν κάποιες συνέργειες. Δεν κοιτάμε τόσο πολύ τις συνέργειες αλλά και την συμπληρωματικότητα. Πρέπει να παραμείνουν διαφορετικά αυτά τα μέσα αλλά ο συνδυασμός πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός και συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να βελτιώσουμε τις ε, συνέργειες και την συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων. Για την παρουσίαση του κ. Φανχάλη. Δεν υπάρχει μόνο διπλή αποστολή, υπάρχει τριπλή αποστολή πέρα από τις επενδύσεις ε, να δημιουργηθούν κάποιες ικανότητες ε, και να γίνουν, όπως είπαμε, να γίνει τη σωστή χρήση αυτών των επενδύσεων. Και όπως είπε ο κ. Φανίσελ, Νομίζω πως αυτή η επιμερισμένη διαχείριση ε, είναι αποτελεσματική σε αυτό το μέτωπο και θα συνεχίσουμε με αυτό το καθεστώς και στο μέλλον. Μετά υπήρχε κάτι άλλο. Ναι, το τελευταίο σχόλιο που ήθελα να κάνω. Γεγονό είναι πως υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί αργήσαμε να εγκρίνουμε τον κανονισμό, αλλά και γιατί υπήρχαν κάποιες καινοτομίες στους νέους αυτούς ε, κανονισμούς και είναι σοβαρές αυτές οι καθυστερήσεις, το βλέπουμε με την αιρεσιμότητα εξ με τη θεματική συγκέντρωση. Δεν θα έλεγα πως ε, είναι θέμα κριτικής, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει, να προετοιμαστούμε καλύτερα και δεν πρέπει να αφήσουμε εκτός όλες αυτές οι μεγάλες βελτιώσεις της πολιτικής μας που πετύχαμε στον νέο κανονισμό, αλλά γεγονός είναι πως ε, Υπάρχουν καθυστερήσεις ε, με τις ε, καινοτομίες, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στα κράτη-μέλη. Και δεν έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της υπόθεσης. Τα έχουμε αιτήσιες ε, διαδικασίες απολογισμού και βεβαίως έχουμε και το νέο πλαίσιο το οποίο θα ξεκινήσει το 2017 με τον έλεγχο με τα λεγόμενα ορόσημα. Αυτό λοιπόν το σύντομο σχόλιο από εμάς ε, και πραγματικά σας ευχαριστώ για την συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλατε να αντιδράσετε κυρίες και κύριοι και με ποια σειρά. Κύριε Φανζάκ. Ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω ορισμένες από τις ερωτήσεις ερώτηση του κυρίου Βανίστεν Ρόι. Έχει δίκιο ότι δεν βλέπουμε πολλές από τις δυνατότητες που δίνονται στο σχεδιασμό των περιφερειακών ε, προγραμμάτων. Δηλαδή βλέπουμε περισσότερους δικαιούχους ή οφειλέτες από άλλα ε, προγράμματα ε, εθνικά ενδεχομένως και όχι περιφαριακές συνεργασίες. Η πραγματική περιφερειακή συνεργασία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί, δεν έχω όμως αναλύσει ακόμα το θέμα αυτό. Ίσως κάποια στοιχεία ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα προγράμματα αυτά δεν είναι γνωστά, δεν υπάρχουν εμπόδια ιδιαίτερα. Ε, επίσης ε, το 15% το οποίο μπορεί να αφορά ε, περιοχές εκτός της ε, επικρατείας της περιφερείας είναι ένα μεγάλο ποσοστό, πάντως δεν χρησιμοποιούνται ακόμα οι διεθνείς σχέσεις στα προγράμματά μας. Ο κ. Βανιστερόη ρώτησε τι γίνεται με τα ITIs, με το Κοινωνικό Ταμείο στην, ε, στις κάτω χώρες. Έχουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, για τις τέσσερις μεγάλες ε, πόλεις οι οποίες έλαβαν ε, κάποια χρήματα ως δικαιούχοι του εθνικού προγράμματος και μετά πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ΙΤΑΙΣ μαζί με το, τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε ακριβώς τον ίδιο κανονισμό ούτε τους ίδιους τρόπους Ε, υποβολής ε, εκθέσεων. Αλλά πάντως ε, έχουμε αυτή την ενιαία θηρίδα, μια μικρή ενιαία θηρίδα. Έχουμε τώρα λάβει το, το ποσά για τα δύο χρόνια και μετά ξανά για τα επόμενα δύο χρόνια. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν συνδυασμού έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πάει κανείς σε δύο διαφορετικούς οργανισμούς να απευθυνθεί. Επίσης με ρωτήσατε αν ε, είναι επικίνδυνο να ξεκινούμε με την εξάντε ερεσιμότητα, μήπως ε, δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ε, μέχρι το τέλος του χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα όταν ε, υπάρχει δηλαδή, δηλαδή ε, εάν τα πράγματα δεν προχωρήσουν καλά τότε μπορεί να παίρνει περισσότερο χρόνο η επένδυση και ε, μπορεί να προβληθεί αν όλα πάνε καλά και κάποια επιπλέον χρονική, κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα. αλλά δεν είμαι και γνώστης ιδιαίτερα του θέματος. Κεντρο, κεντρική αποκεντρωμένη, η διοίκηση, επιμερισμένη διαχείριση. Νομίζω ότι για την καινοτομία, την περιφερειακή, ο καλύτερος τρόπος τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε δει ε, στην, ε, στις κατοχώρες είναι από κάτω προς τα πάνω bottom-up και με περιφερειακή συνεργασία γιατί όταν γίνονται εθνικές ε, ε, προσκλήσεις και διαγωνισμοί τότε βλέπουμε ότι ε, παραμένει, όταν είναι κεντρική η διαχείριση, οι εμπειρίες δεν είναι πολλές, ενώ με αποκεντρωμένη και διαχείριση τότε έχουμε συμμετοχή. Αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Χέλη. Ευχαριστώ. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και παρατηρήσεις έγιναν. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Έχω και αεροπλάνο που πρέπει να προλάβω. Κάποιες παρατηρήσεις λοιπόν. Πρώτον, η φύση της πολιτικής συνοχής. Τι είναι ουσιαστικά. Πρέπει να καταστεί σαφές και σε αρκετές περιπτώσεις νομίζω ότι δεν είναι δώρο η πολιτική συνοχή. Δεν είναι κάποια αντιστάθμιση για το άνοιγμα αγορών. Είναι μια επένδυση στις ίδιες τις χώρες μας, στα κράτη-μέλη και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε κάποια μέτωπα, σε κάποιες πολιτικές συζητήσεις χαίρομαι για το ότι ίδια οι ίδιες οι αλήθειες αυτές που αμφισβητούνται και πρέπει να απαντήσουμε εμεί. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι στην Ευρώπη να θεωρούν την πολιτική συνοχή ε, ως ένα σωρό λεφτά χωρίς ε, να συμμετέχει στους όρους και προϋποθέσεις. Ε, πρέπει λοιπόν να διεξαχθεί αυτή η αντιπαράθεση και να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Βλέποντας διαφημίσεις για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και την ε, στρεβλή παρουσίαση σαν να ήταν μια επένδυση κυβερνητική. Λυπούμε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι κυβερνητική επένδυση. Σε, σε πολλές χώρες μας υπάρχει ένα γράφημα που λέει ότι 60, 70, 80% των ε, ε κονδυλίων που επενδύουν προέρχονται από την Ευρώπη. Μέσα στο πλαίσιο της ε, συγχρηματοδότησης πρέπει να δούμε τον ρόλο και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δική μου τη χώρα η συζήτηση διεξάγεται ε, ως προς το ότι θα ήταν μηδενικό το ποσοστό ανάπτυξης αν δεν είχαμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τι γίνεται όταν βλέπω τις ε, βραδινές ειδήσει, ούτε κουβέντα ούτε λόγος για την Ευρώπη που έχει τόσο σημαντικό ρόλο. Έχουμε εδώ λοιπόν πρόκληση για τις ίδιες τις τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής συνοχής και τις αρχές της Ευρώπης που πρέπει να προασπίσουμε και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και αυτό είναι ένα θέμα για την πολιτική συνοχής που έχει τεράστια σημασία. Δεύτερο, απλούστευση, απλοποίηση ως ίσως σε αντίφαση με την ε, εταιρική σχέση και την ε, πολυεπίπεδη παρέμβαση. Κανένας από εμά δεν είπε, δεν έκανε λόγο για την απλούστευση λέγοντας ότι πρέπει να καταργηθούν οι εποπτικές επιτροπές ή ε, η εταιρική σχέση ή η συμμετοχή των περιφερειών. Πάντα ήμουν υπέρμαχος της περιφερειακής προσέγγισης λόγω της πολυεπίπεδης διαχείρισης και διακυβέρνησης. Και μπορώ να σας πω ότι όταν δημιουργήσαμε την πρώτη Εποπτική Επιτροπή το 2004 για το, τα πρώτα προγράμματα των διαθροτικών ταμείων που λειτουργήσαν. Είχαμε τις οργανώσεις της κοινωνίας ε, των πολιτών που ε, δεν θεωρήσαμε ούτε μπορέσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά. Έγινε δεύτερη φύση μας αυτό και η παρακολούθηση και η εποπτεία δεν νομίζω ότι κανείς όταν κάνουμε λόγο για απλούστευση θα ήθελε να ξεφορτωθεί και να καταργήσει τα στοιχεία αυτά εποπτείας, παρακολούθησης, λογοδοσίας. Αλλά και πάλι με όλο το σεβασμό για τα διάφορα συντάγματα και συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών πρέπει να επιμείνουμε και να εμείνουμε στην πολυεπίπεδη διαχείριση και λογοδότηση και διακυβέρνηση ώστε για να υπάρξει η αηφορία στην, ε, στις πόλεις υπάρχουν δυνατότητες να εμπλακούν οι πόλεις και οι περιφέρειες και οι περιοχές της υπαίθρου ε, και μπορεί αυτό να δημιουργήσει ένα δυναμικό για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ας το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το δυναμικό. Δεν το κάνουν όλες οι χώρες. Υπάρχουν και στοιχεία όπως το ITI που ε, δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και δεν το έχουμε αυτό Στη δική μου χώρα βλέπω μια οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο δεν με ικανοποιεί καθόλου έτσι όπως έχει εξελιχθεί για την υλοποίηση και την εφαρμογή κονδυλίων και την απορροφητικότητα που έγινε σε μια παρέμβαση, τέθηκε αυτή η ερώτηση. Ναι, αληθεύει ότι το πολιετές, ο πολιτής προγραμματισμός από πλευράς ε, προϋπολογισμού είναι πάντα ένα από τα στοιχεία της ε, δημόσιας ε, διαχείρισης και υπάρχουν προβλήματα και στις χώρες των Βαλκανίων είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζεται όμως, βρίσκεται υπό έλεγχο. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση ότι πρέπει να γίνει σωστά ο προγραμματισμός και η διαχείριση και ο καλύτερος τρόπος είναι ο προγραμματισμός για τις ε, δημόσιες επενδύσεις όπως ακριβώς και για την πολιτική συνοχή. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε διαφορετικά με οποιοδήποτε άλλο σύστημα προϋπολογιστικό. Το χειρότερο σενάριο μπορεί να είναι ορίστε αυτά είναι τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας αλλά έχουμε πολιετής δεσμεύσεις και κονδύλια υποχρεώσεων και πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε υπό αυτούς τους περιορισμούς. Μια και το, τους υπουργούς και τα υπουργεία μπορούν να τα, βοηθήσουν οι επενδύσεις αυτές. Δεν μπορεί να θέλουμε να, εξοικονομ... να, να διασφαλίσουμε αυτά τα κονδύλια ώστε να χρησιμοποιηθούν σε μια υστερότερη φάση. Γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε επιστροφή και πρόσθετη αξία. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τα επενδύσουμε σωστά και και και για να δούμε και την απορροφητικότητα στο τέλος τέλος όταν βλέπουμε ότι υπάρχει διασπάθηση κονδυλίων ή μη αποτελεσματικότητα υπάρχουν α, τροτά σημεία, ευάλωτα σημεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επανορθωθούν. Δεν είναι κάτι το ανέφικτο να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί η κύρια παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα προγράμματα από ότι ε, τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα. Δεν πρέπει λοιπόν εδώ να φοβούμαστε να επιμένουμε και να εμένουμε σε κάποιες αρχές. Ευχαριστώ. Θα θέλετε να απαντήσετε κι εσείς, κυρία μου. Ναι, αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την ε, δικιά μου παρέμβαση πρώτο σχετικά με τις ε, εταιρικέ ε, συμφωνίες. Εδώ βλέπουμε ότι έχει υπάρξει πρόοδος ε, και τώρα πλέον μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, ε, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για το κλίμα και την ενέργεια. ενδεχομένω, βέβαια δεν πρέπει να είμαστε και υπερβολικά ενθουσιώδεις γιατί θα πρέπει αυτή η δυνατότητα παρέμβαση να ακολουθηθεί και από ε, συγκεκριμένες δράσεις. Ε, πάντως, ε, σίγουρα ένα καλό βήμα είναι αυτές οι συμφωνίες εταιρική σχέσης. Κάτι άλλο, διεθνής χωρική συνεργασία, τα προγράμματα περιβαλλοντικής συνεργασίας ε, είναι σημαντικά, εξαρτάται βέβαια και ποιος είναι ο στόχος που βάζει κανείς. Για να σας δώσω ένα ε, παράδειγμα, ε, υπάρχει τώρα στα Σκαριά ένα σχέδιο για τον Δούναβη, όλες οι χώρες, οι παραδουνάβιες, οι οποίες θα συνεργαστούν γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις οτιδήποτε κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες σε μία περιοχή έχει επίπτωση σε μια άλλη ε, περιοχή των ε, παραδουνάβιων ε, χωρών. Επομένως, οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, να υπάρχει συνεργασία, οι στόχοι να είναι μετρήσιμοι και να γίνονται σε διεθνές περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γκορέζο. Κοιτάξτε, η προσέγγιση αυτή των επενδύσεων έχει το εξή πρόβλημα σε τι θα πρέπει να επενδύσουμε στην ικανοποίηση των πολιτών ή στην μελλοντική ανταγωνιστικότητα και την θέση μας στην παγκόσμια οικονομία. Μέχρι τώρα εμείς ε, στο δικό μας μέρος της Ευρώπης επενδύουμε περισσότερο στο να ικανοποιήσουμε τους πολίτες παρά στη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Διακρίνουμε βεβαίως μεταξύ της ενίσχυσης της ε, ζήτησης ε, που είναι προσωρινή αλλά εμφανής ε, και την ενίσχυση της προσφοράς που θα ωφελήσει γενικότερα την οικονομική αποτελεσματικότητα του συστήματος παραγωγής. Από μακροοικονομικές και μικροοικονομικές μελέτες βλέπουμε ξεκάθαρα πως η ενίσχυση της ζήτησης μέχρι στιγμής είναι πολύ ισχυρότερη από ότι της ε, προσφοράς. Οπότε ικανοποιούμε τον πληθυσμό, έχουμε ανάπτυξη, σχολεία, ε, πάρκα κτλ. Αλλά δεν έχουμε καινοτομία, δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα. Εάν μιλάμε λοιπόν για καινοτομία, και εδώ πέρα πάει η παγίδα των χωρών μέσου εισοδήματος, ε, βλέπουμε πως μέχρι ένα επίπεδο ανάπτυξης είναι αποτελεσματικό το ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά από ένα επίπεδο και μετά είναι αποτελεσματικό το κοινωνικό κεφάλαιο. Δεν είναι λοιπόν ότι αυτοί που διαχειρίζονται τα λεφτά δεν ε, ε, εμπιστεύονται τους ε, καινοτόμους ή αν ο επιχειρηματίας δεν εμπιστεύεται τον επιστήμονα. Αν ο επιστήμονας δεν εμπιστεύεται αυτόν ο οποίος θα κάνει την ε, καινοτομία δεν Δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις δικές μας τις χώρες και πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη στη δημόσια σφαίρα και μεταξύ αυτής και της σφαίρας έρευνας και ανάπτυξης και των επιχειρηματιών. Και υπάρχει μια τάση και μια αποδοχή του ρίσκου. Χωρίς, χωρίς ρίσκο δεν υπάρχει καινοτομία και μπορούμε να δούμε αυτούς που χρηματοδοτούν καινοτόμα έργα φοβούνται ε, τον κίνδυνο όπως ο διάολος τον, τον αγιασμό. Ε, δεν γίνεται αυτό όμως. Μετά, αξιολογιστή αξιολογούμε. Αξιολογούμε τις δραστηριότητες μας για να τις ε, βελτιώσουμε ή για να ικανοποιηθούμε ότι τα κάναμε όλα σωστά και να αποδείξουμε και στους έξω ότι είμαστε αποτελεσματικοί. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά οι αξιολογήσει είναι κατακαιρματισμένες, ε, τυπικές και γίνονται απλά για να λέμε ότι τα πήγαμε καλά. Και για να αποδείξουμε και στους έξω ότι είμαστε αποτελεσματικοί για να υπερασπιστούμε δηλαδή την πολιτική μας για τους ανταγωνιστές ε, που θέλουν και αυτοί το μερίδιό τους από τα κονδύλια της συνοχής. Και βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ότι αυτοί οι οποίοι χαράζουν στρατηγική σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο περιφερειακό επίπεδο συχνά βλέπουμε ότι τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα είναι σημαντικότερα από την ε, αναπτυξιακή στρατηγική, ενώ πρέπει να σημαίνει το αντίστροφο. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια λοιπόν διαμορφώνουν το πώς σκεφτόμαστε για το μέλλον μας και οι προτεραιότητες και οι πολιτικές ε, της Ένωσης διαμορφώνουν την στρατηγική μας ε, σκέψη. Πρέπει να θυμόμαστε πως ε, πολλά λεφτά πάνε στην κέντρο-ανατολική Ευρώπη, αλλά είναι τι να σου πω, ένα 10-15% των, των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι 50-60-70% των δημοσίων επενδύσεων. Αλλά οι επενδύσεις που γίνονται στην οικονομία, στην ανάπτυξη, ε, είναι πολύ χαμηλή και λέω συχνά στη χώρα μου πως τα κονδύλια της συνοχής δεν θα μας σώσουν. Μόνοι μας πρέπει να σωθούμε. Πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί, ε, έξυπνοι, καινοτόμοι, η χώρα μας στο μέλλον και στην Νότια Ευρώπη το ίδιο. Ίσως και στην Ευρώπη συνολικά. Είναι μια ωραία ήπειρο, αλλά όχι τόσο αποτελεσματική όσο άλλες ήπειροι. Και αυτή είναι η πρόκληση για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις των πραγματογνωμόνων μας που ήταν πάρα πολύ γόνιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε με τη συζήτηση για την απουσία εμπιστοσύνης. Αυτό έγινε όταν ξεκίνησε η συζήτηση του πιθανού μέλλον, ε, δυνάμει μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε αυτό το στοιχείο της απουσίας εμπιστοσύνης μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών, μεταξύ των ε, ε, διαχειριστικών αρχών, μεταξύ των εποφελούμενων ε, αποδεκτών και τέλος μεταξύ των ίδιων των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Απουσία εμπιστοσύνης. Με εξέπληξε να το ακούσω από εσά κύριε Γκοζέλα αυτό το ίδιο θέμα. Απουσία έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό το θέμα της έλλειψης απουσίας εμπιστοσύνης. Είναι το αίτιο και η βάση για να υπάρξει και να δημιουργηθεί αυτή η επικοδόμηση, αυτό το επικοδόμημα για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα λάβουν τον λόγο οι συγητές. Τώρα ο κύριος Πυρίνσκι πρώτος. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Και πάλι ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις που έγιναν από τους πραγματογνώμονες και τις τοποθετήσεις τους. Επανερχόμενος τώρα στο έγγραφο το οποίο είναι υποσυζήτηση την ανακοίνωση δηλαδή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πω ότι το άρθρο 16 κάνει λόγο για την προπαρασκευή μιας μελέτης, σύνταξη μιας μελέτης και την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούμε ότι αυτή η ανακοίνωση είναι το θέμα αυτής της έκθεσης. Δεν είμαι όμως βέβαιος αν αυτές οι δύο έννοιες ή προσεγγίσεις, αυτές, αυτοί οι δύο όροι ταυτίζονται στην ίδια την πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με το τι παράγεται ε, και τεκμηριώνεται. Αλλά πιο σημαντικό ακόμα είναι τι είναι αυτό το οποίο ερμηνεύουμε υπό τον τίτλο αυτής της ανακοίνωσης και πώς το βλέπουμε. Λέει, επενδύσεις στην ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, μεγιστοποιώντας επενδύσεις από πλευράς Ευρωπαϊκών Διαθωτικών Ταμείων και ήδη τέθηκε το ερώτημα, συνεισφορά προς τι, προς ποιο σκοπό. Διότι στο δημοσίευμα τύπου Δεκεμβρίου 2014 στην ανακοίνωση τύπου η συνεισφορά αυτή ήδη θεωρείται ως συνεισφορά των διαθροτικών και επενδυτικών ταμείων στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι ότου καταλήξουμε στο τελικό νόημα και εγχείρημα αυτών των ε, συμφωνιών εταιρικής σχέσης και σε τι στοχεύουν και τι υποτίθεται ότι θα επιτύχουν. Και εδώ ερχόμαστε στο θέμα το οποίο ανέφερα για το τι συζητούμε, τι βρίσκεται υποσυζήτηση, περί τίνος πρόκειται. Συνοχή, ή τρίτη έννοια, η προσέγγιση προπαρασκευής ενός μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αυτών. Είναι ζωτική σημασία, Πρόεδρε, να προσαφηνήσουμε για ποιο πράγμα κάνουμε λόγο εδώ. Κάνουμε λόγο για τα διαδροτικά ταμεία που υποτίθεται ότι θα εξυπηρετήσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ίδια την Ένωση. Είναι λοιπόν συνοχή μεταξύ περιφερειών αυτή η συνοχή. Και το άρθρο 174 της ε, ε, Ένωσης τι λέει για την ε, συνεργασία, συνοχή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ανισότητες σε σχέση με το επίπεδο ανάπτυξης των διαφορετικών περιοχών και την ε, ε, μειονεκτικότητα των λιγότερο ευνοημένων περιοχών πρέπει να τις χρησιμοποιήσει ως σημεία αναφοράς. Μπορούμε να κάνουμε λόγο λοιπόν για τις επενδύσεις υπό διαφορετικά κεφάλαια και έννοιες. Αλλά να είμαστε σαφείς, όταν κάνουμε λόγο για διαθωτικά ταμεία, κάνουμε λόγο για επενδύσεις στην συνοχή και στις δραστηριότητες και δράσεις υπέρ της συνοχής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εδώ δεν είναι φυσικά κάτι το ο, οτιδήποτε, είναι επενδύσεις, στο τέλος τέλος όμως είναι επενδύσεις στην ίδια την Ένωση. Δηλαδή για μια πιο εναρμονισμένη ανάπτυξη, πιο αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην ανακοίνωση υπάρχει το επιχείρημα και αναφέρεται ότι η κρίση διέγραψε και ε, ε, εξέλιψε όλα αυτά ε, τα κέρδη και τα ωφέλη σε σχέση με τα κράτη-μέλη από το 2000. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι πώς αυτές οι εταιρικέ σχέσεις και τα λειτουργικά προγράμματα για την περίοδο 2009-2014 ήταν αρκετά θετικά στοχευμένα για να ανακτηθεί η σύγκληση και η συνοχή. Ε, έχουμε συνειδητοποιήσει τις αυξημένες διαφορές και τις παρεκκλήσεις και γίνονται επενδύσεις με τέτοιο στοχοθετημένο τρόπο ώστε να μπορεί να υπάρξει συνδιαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ώστε τα τελικά αποτελέσματα να είναι πραγματικά αυτά τα οποία επιθυμούμε και να είναι υποφελή και βλέποντας εδώ την παρέκκληση που υπάρχει με τους μέσους όρους όσον αφορά τα, το στοιχείο του ΑΕΠ για το 2013 για παράδειγμα Νομίζω δεν υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με το 2009. Ίσως μάλιστα υπάρχει και κάποια επιδίνωση ακόμα περισσότερο και όχι πρόοδος. Όταν κάνουμε λόγο λοιπόν για τη συνεισφορά των διαθωτικών ταμείων τελικά ως αποτέλεσμα, έχει τεράστια σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να εξισώσουμε αυτή τη συνεισφορά με την πραγματικότητα που αναφέρεται στη σελίδα 2 όσον αφορά τις προτεραιότητες της ε, νέας Επιτροπής. Ψηφιακή ε, ε, εποχή, ψηφιοποίηση, ψηφιακή Ευρώπη και όλων των προτεραιοτήτων με συγκεκριμένες συστάσεις όπως διατυπώνονται. Αυτά δεν στοχεύουν στην κατεύθυνση που πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να έχουμε απόλυτα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να είναι η κύρια ανησυχία μας και το μέλημά μας για αυτές τις χώρες και για τα διαθωτικά ταμεία. Θα πρέπει λοιπόν να μην τα περιπλέκουμε υπερβολικά τα πράγματα. Κάνουμε απλά λόγο για απασχόληση, για θέσεις απασχόλησης, για ανάπτυξη, για ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, ποιότητα διαβίωσης, ε, αναβάθμιση της ποιότητας ε, και όλα αυτά είναι αυτά τα οποία αναμένουμε και θα έπρεπε να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να στοχεύσει προς την επίτευξή τους. Ελπίζω ότι ο, πρόεδρος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής θα διαβιβάσει αυτή την παρατήρησή μου στην Επιτροπή και να ληφθεί αυτή η υπόψη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φανίστερ Ρό, είχε τον λόγο για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πολύ με τον συνάδελφο από την Επιτροπή Απασχόληση, γιατί ξέρετε για την ανάπτυξη και τις δουλειές. Αυτό είναι μόνο ένας από τους στόχους που έχουμε όταν είχαμε ακριβώ και την θεματική επικέντρωση για το 2014 με 20 πρόκειται για μια επαναδιατύπωση όσων είχαμε συμφωνήσει στον νέο κανονισμό στην περίοδο αυτή. Όλα αυτά λοιπόν αναδιατυπώνονται στις νέες προτεραιότητες της Κομισιόν. Δηλαδή μιλάμε για αηφορία, για τις τέσσερις θεματικές ενότητες είναι κάτι ευρύτερο. Πώς θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά τα οποία μας παρουσίασε η Κομισιόν. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τα όσα ζητήσαμε τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, η τοπική εταιρεία, αν έγιναν. Υπάρχει λοιπόν μια κάποια ε, ένταση θα έλεγα. Δηλαδή θεωρητικά και εγώ έχω τις ίδιες ερωτήσεις ε, αλλά από την άλλη, όταν μιλάμε για συνοχή, η συνοχή στις τρεις αυτές ε, διαστάσεις είναι ένας ξεκάθαρος στόχος της Ένωσης είναι στις συνθήκες, οπότε δεν εκτάμε την συνοχή ως ε, επένδυση ή ως μια διαφοροποιημένη πολιτική. Μπορούμε να πούμε το, το εξής, ότι θα πρέπει να γίνει αυτό και σε σχέση με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση ή τον προσανατολισμό της νέας πολιτικής. Θεωρώ λοιπόν πως έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία σε αυτή την έκθεση να συνεργαστούμε με τα μέλη των επιτροπών μας για το τι θα γίνει στο μέλλον. Και νομίζω πως η σημερινή ακρόαση μας ε, ανέπτυξε τις διαφορετικές απόψεις για το που πηγαίνουμε. Δεν είναι μόνο θέμα λοιπόν ε, ένας προϋπολογισμός για κάποιες αποζημιώσεις, είναι θέμα διαφορετήσεις για να μπορέσουν οι πολίτες μας και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι να βρεθούν σε μια διαφορετική αφετηρία και μετά να υπάρξει μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία στο κέντρο των όσων κάνουμε. Αυτό είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Το θύμενε λοιπόν είναι πάρα πολύ θετικό. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και νομίζω πως υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον ε, και από τους βουλευτές και τους κοιόδης για να το συζητήσουν τώρα. Κοιτώντας πιο λεπτόμερος ε, τα πράγματα, χαίρομαι για το ότι Έχουμε εδώ πέρα τα βασικά τεχνικά στοιχεία των όσων παρουσιαστεί. Η θεματική εστίαση, τα κριτήρια αποτελεσματικότητας, Θα μπορούσαμε έτσι να προσαρμόσουμε το σκεπτικό αυτό. Π.χ εμείς συμφωνήσαμε να πάμε σε έναν προπολογισμό με βάση τα αποτελέσματα. έτσι ως μια μαγική λέξη. Είμαστε λοιπόν τώρα στη μέση της διαδικασίας και έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν συζητάμε ξαφνικά αν πηγαίνουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Και γεγονό είναι ότι μιλάμε για τις εκθέσεις εφαρμογής. Υπάρχουν επίσης κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Γιατί εάν χρησιμοποιήσουμε τα ταλέντα που υπάρχουν, τα κονδύλια πρέπει να εξοδευτούν με τρόπο πολύ αποτελεσματικό και δεν μπορούμε να επανεφεύρουμε τον τροχό. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν αυτή η ε, διαπεριφερειακή συνεργασία με προβληματίζει. Γιατί εάν δεν ε, βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος απόδοσης. Αλλά νομίζω μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω ε, θα είναι πιο αποτελεσματική από το παρελθόν και υπάρχει και λόγος να γίνει αυτή η σύνδεση με τις προτεραιότητες της Κομισιόν που αναφέρατε. Πώς θα προσαρμοστούμε λοιπόν στους στόχους αυτούς για να δείξουμε κάποια αποτελέσματα. Και μία τελευταία παρατήρηση γιατί οπωσδήποτε θα γίνουν και άλλες συζητήσεις ε, τον Ιούλιο κιόλας και θα παρουσιάσω και εγώ ένα έγγραφο με κάποια σημεία κλειδιά και το Σεπτέμβριο μετά τις διακοπές θα έχουμε το πρώτο σχέδιο έκθεσης το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος, ο συνάδελφος από την Ουγγαρία. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός να πούμε δηλαδή ότι ναι τώρα συνεργαζόμαστε σε ένα έργο. Όχι δεν υπάρχει αυτό. Και δεν το βλέπω πουθενά. Και οι πολίτες μας ε, δεν ε, το αντιλαμβάνονται. Εάν οι κυβερνήσεις μας, οι συμπατριώτες μας στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν επικοινωνούν. Ίσως σε κάποια πράγματα όπως ορίζοντας 2020 υπάρχουν κάποια σημεία όπως οι βασικές ε, τεχνολογίες την περιφερειά μου για την τεχνολογία που αναπτύσσεται και όλα αυτά μπορούμε να τα κρατήσουμε στην Ευρώπη π.χ. την Airbus εντάξει μπορούμε να πούμε ότι η Airbus ε, φτιάχνει σε διάφορες χώρες ε, κομμάτια αλλά αν είμαστε αν δεν ήμασταν ενωμένοι θα χάναμε αυτή την δυνατότητα γιατί αν δεν το χρησιμοποιήσουμε θα το χάσουμε δηλαδή και μετά πουλάμε ξέρω εγώ χιλιά Airbus ε, σε δύο χρόνια και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε λοιπόν π.χ. ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ότι πουλήσαμε περισσότερα Airbus από Boeing. Εντάξει, μπορούμε να μοιράσουμε τα λεφτά σε όλους. Όχι, δεν είναι σωστό όμως. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την εδαφική πτυχή, για κάποια στόχευση. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει για να πείσουμε σας ασκούν κριτική στην πολιτική μας να γίνει μια σωστή συζήτηση π.χ. για το Ταμείο Χιούνκερ. Θέλεις. Ε, οπότε εξυπηρετούμε τους στόχους ε, της ε, συνοχής για να εξυπηρετηθούν και σε μια, νέο, σε μια νέα περίοδο που χρειαζόμαστε όλα τα ταλέντα. Στα επόμενα 40 χρόνια η Ευρώπη θα καταλήξει να έχει δύο συνταξιούχους για κάθε εργαζόμενο. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτική η οποία θα μας δώσει δυνατότητες. Και άκουσα πολλές λέξεις που έμαθα από σας σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ε, ειδικού ε, που ακούσαμε και είμαι πεπισμένος ότι από κοινού θα έχουμε μια πιστική έκθεση και θα πείσουμε τους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν ίσως ε, τώρα τόσο καλά την πολιτική της συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή η ακρόαση που κάναμε σήμερα μας έδωσε πολλά νέα εργαλεία και γνώσεις για την επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συμμετείχαν. Ολοκληρώνεται η διαδικασία μας, η συνεδρίασή μας για σήμερα. Η Πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς. Αύριο 9 η ώρα παρακαλώ.